Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι είσαστε εδώ παρόντες και όσοι συμμετέχοντες είναι εξ αποστάσεως. Κάποιες τεχνικές ανακοινώσεις. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Interactio για τις εξαποστάσεων συνεδριάσεις. Γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ουγγρικά, πολωνικά και σλοβενικά είναι οι γλώσσες που, ε, για τις οποίες έχουμε διερμηνία και παθητικά, λιθουανικά και ρουμανικά. Μόνο οι ενεργώς ε, συμμετέχοντες ε, που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών μπορούν να πάρουν το λόγο. Αυθόρμητες αντιδράσεις δεν επιτρέπονται. Παρακαλούμε να έχετε στο κλειστό το μικρόφωνο σας όταν δεν ε, μιλάτε για να μην έχετε δε αντίχηση, καλό να χρησιμοποιήσετε ακουστικά. Θα πρέπει να προσθέσετε το πλήρες όνομά σας όταν θα, συνδεθείτε για να μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε. Οι παθητικοί συμμετέχοντες μπορούν να βάλουν ε, στο listening mode ή να παρακολουθούμε web streaming τη συνεδρίαση και εάν δεν είναι καλή η σύνδεση μπορούν να αποσυνδεθούν και να περάσουν στο web streaming. Θα ψηφίσουμε τώρα το σχέδιο έκθεση ισχυρή Κοινωνική Ευρώπη για τη δίκαιη μετάβαση. Γνωρίζετε ότι είμαστε από τι πρώτε επιτροπέ που άρχισαμε να χρησιμοποιούμε το νέο σύστημα ηλεκτρονική ψηφοφορία EP Vote, που θα το χρησιμοποιούν όλε οι επιτροπέ μέχρι τα τέλη του τρέχοντο. Σήμερα λοιπόν θα ψηφίσουμε το σχέδιο έκθεση όπως σας είπα μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για τη δική μετάβαση. Θέλω να ευχαριστήσω την γραμματεία μας γιατί εργάστηκε κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση χρόνου για να προετοιμάσει τον κατάλογο ψηφοφορία. Τη Μίνα, την Μπάρμπαρα και την Ελοντή. Σας ευχαριστώ πολύ νυχθημερών και μέχρι και το Σαββατοκύριακο εργάστηκαν για να είναι όλα έτοιμα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν έχουμε πολύ προσωπικό στη διάθεσή μας ε, τώρα που προετοιμάζουμε τι εργασίε μας και όλες οι ομάδες θα πρέπει να σέβονται και να τηρούν όλες τις προθεσμίες ανεξαρτήτως ε, ε, πιέσεων μπορεί να υπάρχουν για να αντιμετωπιστεί αυτή η έλλειψη προσωπικού και να μην έχουμε προβλήματα. Θα σας εξηγήσω τώρα πώς ε, μπορούμε να ψηφίσουμε. Έχετε ήδη λάβει βαθμιδών τις οδηγίες για τα διάφορα βήματα που θα πρέπει να κάνετε, πώς θα υποβάλλετε τα ψηφοδέλτιά σας. Ε, η πρώτη ψηφοφορία, τροπολογίες από τις 4 και 45 έως τις 6:30 θα μπορείτε να ψηφίσετε. Όταν ξεκινήσει η θα λάβετε email από το γνωστό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Θα πάρετε το link και για το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσο είναι ανοιχτή ψηφοφορία θα πρέπει να επιλέξετε ηλεκτρονικά στο e του τι θα ψηφίσετε, μετά να ε, φτιάξετε ένα PDF ψηφοδέλτιο που θα πρέπει να στείλετε στο amplevote.europarl.europa.eu ε, από τη δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση εφόσον ε, αρχίσει η ψηφοφορία και όχι αργότερα από τις 6.30. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το ε, IT support ε, για τους βουλευτές. Τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας ε, θα ανακοινωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα. Και στο δεύτερο γύρο που θα έχουμε τις τελικές ψηφοφορίες, αύριο 3η 17 Νοεμβρίου, μπορείτε να ψηφίσετε από τις 11.30 έως τις 12.15. Επίσης, θα ανακοινωθεί με email ημερομηνία και ώρα μάλλον έναρξη και λήξης της ε, ψηφοφορίας. Και η ίδια διαδικασία θα ισχύει όπως ε, και για αυτή την ψηφοφορία μέσω του EP Vote. Ε, θα ελέγξουμε τώρα για την πρώτη ψηφοφορία αν έχουμε απαρτία. Πώς πηγαίνουμε, πόσα μέλη είναι στα δεδομένα, πόσοι βουλευτές. Παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί που λέει Raise Hand. Ωραία, πηγαίνουν πολύ καλά από ό,τι φαίνεται. Ωραία, ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν απαρτία. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 5 που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μάικλο Φλάχερ, τη Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με τα πορίσματα του οργανισμού όσον αφορά τους Ρωμά και τους πλανοφίους κατά την πανδημία και όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένου κατά την πανδημία. Πρέπει, πρέπει, to stop the spread of the virus and avoid για να μην επιβαρυνθεί το σύστημα υγείας. Ε, υπάρχουν μέτρα ε, και έχουν σίγουρα επηρεάσει όλα αυτά θεμελιώδη δικαιώματα πολλών ομάδων, ιδίως ευάλωτων ομάδων και κάποιες ομάδες μάλιστα έχουν πληγεί δυσανάλογα σε σχέση με άλλους. Ε, υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης, κίνδυνος όμως απομόνωσης λόγω του περιορισμού επαφών ιδίως για τους ηλικιωμένους ε, στους οίκους ευγυρίας. Αλλά και τα άτομα με αναπηρία έζησαν ε, τις ε, διαταραχές αυτές στην παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης. Οι Ρώμα, οι επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας λόγω του συνοστισμού, λόγω του τρόπου διαβίωσής τους. Θα να ε, καλωσορίσω και την Ελένα Ντάλη, την Επίτροπο, η οποία θα παρακολουθήσει την ανταλλαγή απόψεων αυτή. Θα καλωσορίσω και τον Μάγκλο Φλάχερτη, που είναι ο Διευθυντή του Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για τρία λεπτά θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επίτροπο, την κυρία Ντάλη, και εν συνεχεία στον ε, κύριο Διευθυντή, ε, τον κύριο Φλάχερτη, για το ΦΡΑ. Παρακαλώ, κυρία Ντάλη, έχετε το λόγο για τρία έως πέντε λεπτά. Madame Dali, please press the speak button. Είστε το κουμπί του μικροφώνου, το speak, το speak, λέει ο γραμματέας στην κυρία Ντάλη. Με ακούτε, λέει η κυρία Ντάλη. Ναι, αλλά δεν σας βλέπουμε. Oh. You connect your video, please. Πρέπει να συνδέσετε και την εικόνα, το βίντεο. Τώρα με βλέπετε, λέει κύριε Αντάλη. Μάλιστα, μάλιστα, μιλήστε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στη σημερινή συζήτηση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, θα έχουν επιπτώσεις. Πρόκειται για πάρα πολύ ευάλωτους, για μειονεκτούντες. Είναι ε, αυτοί οι άνθρωποι μία από τις προτεραιότητές μας και η σημερινή ε, συζήτηση θα βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά μας. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντική Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυσμενείς διακρίσεις, κοινωνικός αποκλεισμός. Όλα αυτά είναι μια κοινωνική πραγματικότητα. Έχουν φύγει πάρα πολλά από όλα αυτά η Ρώμα. Είναι η στέγασή τους πάρα πολύ κακής ποιότητας και με την πανδημία εφήγησαν όσο όσο κανείς άλλος, γιατί έχουν θέματα ε, προσβασιμότητας ε, στην υγιεινή και στις υπόλοιπες κοινοφιλείς υπηρεσίες. Εμείς προσπαθούμε επομένως να εντοπίσουμε ε, τις οικονομικές επιπτώσεις εκτός από τις υγειονομικές, γιατί σε κάποια κράτη οι, οι Ρωμά, τσιγκάνοι Ρωμά, αντιμετωπίζονται ως απειλή για την υγεία, έχουν στιγματιστεί. Ζητάμε συγγνώμη, αλλά είναι πολύ κακό ο ήχο τη κυρία Ντάλη. Ενέκρινε στι 7 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πλαίσιο δράση για τους Ρωμά. Καθορίσαμε τους στόχους μας για τα επόμενα χρόνια για να δούμε ακριβώς πώς θα τους πετύχουμε. Με βάση τις νέες ανάγκες επί τη βάση αυτής της Προτείναμε μία σειρά από χρηματοοικονομικά μέτρα για να τους στηρίξουμε. Και έτσι έχουμε τέτοιους ε, στόχους για συμμετοχή, για ισότητα, υγεία, στέγαση. Όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πόσιμο νερό, και κάτι να γίνει για τις τόσο πυκνοκατοικημένες τους ε, κοινότητες και δήμους. Είναι και το θέμα βέβαια των ανθρώπων με αναπηρία. Ακούμε τους ανθρώπους που στην πράξη ασχολούνται με αυτά τα προβλήματα και προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με την παροχή αυτών των υπηρεσιών και μιλάμε και με τους χρήστες αυτών. Αντιδράσαμε πάρα πολύ γρήγορα για να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε ιατρικό υλικό, προστατευτικό υλικό. Όλα αυτά στα πλαίσια του σχετικού πακέτου για τον COVID. Και θα αξιοποιήσουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο επί τη βάση των όσων προβλέπει ο ΕΕ για τους ανθρώπους με αναπηρία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, να γίνουν κάποιες αλλαγές, να γίνουν επενδύσεις, γιατί χρειάζεται κάτι να κάνουμε και να υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες υποστήριξη αυτών των ανθρώπων εκεί στους Δήμους και που ζουν και όλα αυτά τα προβλήματα που προϋπήρχαν τα ανέδειξε η πανδημία. Στρατηγική για τους ανθρώπους με αναπηρία, να συμπληρώσουμε τις εθνικές στρατηγικές να προστατεύσουμε την υγεία αυτών των ανθρώπων, να έχουν πρόσβαση και αυτοί σε υπηρεσίες υγείας και στην πρόληψη επίσης των προβλημάτων της υγείας. Όλες αυτές οι δυσκολίες έχουν θίξει αυτούς τους ανθρώπους με πολλούς τρόπους. Θα πρέπει να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να απολάβουν όλων των δικαιωμάτων, όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων σύμφωνα με το σχετικό χάρτη. Τώρα χρειάζονται ακόμη περισσότερο από ό,τι προηγουμένω ιατρική φροντίδα, Κοινωνικέ υπηρεσίε. σε καθημερινή βάση. Όπως και οι μεγαλύτεροι των 65, έτσι και οι ανάπηροι υπήρχαν πολλά προβλήματα, χρειαζόταν η προστασία των δικαιωμάτων τους και το 2020, τον Ιούνιο, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι χρειάζεται κάτι να γίνει και θα πρέπει επίσης να καλυφθούν οι ανάγκες ενός γεράσκοντος πληθυσμού πέραν των ανθρώπων με αναπηρία. Βέβαια, όλα αυτά είναι εθνική αρμοδιότητα, αλλά έχουμε εμείς τον κοινωνικό πυλώνα. Οπότε πρέπει ο κόσμος να έχει πρόσβαση σε ποιοτικέ ε, κοινωνικέ υπηρεσίε και εμεί προσπαθούμε να καταλάβουμε πρώτε καλύτερε πρακτικέ, να προσφέρουμε την ευγνωμοσύνη και έτσι να μπορέσουμε να καθισχάσουμε αυτού που είναι ευάλωτοι, όπω οι πιο ηλικιωμένοι, όπω αυτοί με ε, αναπηρία, θα πρέπει, εάν ε, μολυνθούν, θα πρέπει να έχουν τη δέουσα αγωγή σύμφωνα με τα υπάρχοντα αντικειμενικά κριτήρια, οπότε ε, είχαμε την υπηρεσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ήταν ένας ε, πολύτιμος συνεργάτης. Οπότε περιμένω πώς και πώς να ακούσω τι θα πει η κυρία Σοφλάχερτη που θα μας παρουσιάσει ε, τα αποτελέσματα της μελέτης των μελετών της υπηρεσίας του για αυτούς τους ανθρώπους. Με τη σημερινή συζήτηση και εμείς θα καταγράψουμε τη γνώμη σας για αυτές τις στρατηγικές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε την κυρία Νταλή. Ήταν ωραίο που σας είδαμε ακόμα και μόνο στην οθόνη. Θα ακούσουμε τον κύριο Φλάχατσι τώρα, τον Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρέπει να περιμένουμε λίγα λεπτά γιατί έχουμε χάσει την επαφή με τον κύριο Φλάχατη. I ask you Ζητώ την υπομονή σας διότι οι τεχνικοί προσπαθούν να αποκαταστήσουν την επαφή. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε καταφέρει, μέχρι αυτή τη στιγμή δηλαδή. So, unfortunately... Δυστυχώς, λέει η πρόεδρος, φαίνεται ότι δεν, δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε την επαφή με τον κύριο Φλάχετη και επομένως πρέπει να συνεχίσουμε διότι έχουμε και κανόνες σχετικά με το χρόνο στον οποίο διατίθεται διερμηνία. Προτείνω να πάμε στο σημείο 6 αλλά δεν ξέρω κιόλα. Πρέπει να βεβαιωθώ ότι έχουμε όλους αυτούς που πρέπει να έχουμε συνδεδεμένου για να μπορέσουμε να πάμε στο 6. Η κυρία Λάγκεν Ζήπιν, η κυρία Νταλή ε, νομίζω ότι είναι ακόμα συνδεδεμένη. Και για τον πρώτο γύρο ερωτήσεων έχουμε τον κύριο Κώσα. Είναι, είναι Όχι. Ο κύριο Έιντζελ, ο κύριο Άγχελ η κυρία Μάξοβα. Η κυρία Ζαμέ. Ναι. Ντελαπίσα. Ωραία. Περέιρα. Εντάξει. Θα προσπαθήσουμε έτσι. Ε, συνάδελφοι, λοιπόν, καθότι χάσαμε... Α, το ξαναβρήκαμε τον κύριο έτσι. Μόλις μου είπαν οι τεχνικοί, τον έχουμε με καλή σύνδεση και όλα αυτά και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθετε κύριο Φλάιτι στην Επιτροπή Απασχόλησης για πολύ ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν στον οργανισμό σας. Σας δίνει το λόγο. Έχετε 15 λεπτά για να μας παρουσιάσετε τα πορίσματά σας. Παρακαλώ. Αν μπορείτε να πατήσετε το κομβίο του μικροφόνου. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα. Ο Οργανισμός Τεμελιωδών Δικαιωμάτων παρακολουθεί στενά τις ε, πτυχές θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλη αυτή την κρίση πανδημίας. Έχουμε λοιπόν συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των δικαιωμάτων της πανδημίας και αντιδράσεων προς αυτήν στα 27 κράτη-μέλη. Όπως είπε η Επίτροπος και η Πρόεδρος, βλέπουμε πολύ διαφοροποιημένο αντίκτυπο της πανδημίας που πλήττει ευάλωτες ομάδες με πολύ διαφορετικό και ανισόρροπο τρόπο. Η Ρωμά οι άνθρωποι με αναπηρίε και οι πιο ηλικιωμένοι, υπογραμμίζω ήδη. Η κοινότητα των ομάδων και η Ρωμά είναι οι μεγαλύτερες μειονότητες μας. Περί τα 6 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολύ σημαντικά στοιχεία, ανεξαρτήτως του COVID, της ε, περιθωριοποίησής τους ε, και των ε, καταχρήσεων, των διακρίσεων με που υφίστανται και συντάσσουμε και μια έκθεση ανά κράτος μέλος για να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης για το θέμα αυτό. Και πάλι λέω, ανεξαρτήτως του COVID έχουμε ανησυχητικά επίπεδα προσδοκίμου που είναι πολύ χαμηλότερο από του γενικού πληθυσμού, ένδυας, ε, διακρίσεων και μίσους. Όπως η Επίτροπος Ντάλι είπε, όλα αυτά έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες με την κρίση της πανδημίας. Πολλοί Ρωμά και ε, νομάδες βρίσκονται σε, κατέχουν θέσεις απασχόλησης ε, ιδιαίτερα ευάλωτες και που πολλοί, πολλές από αυτές έχουν χαθεί το τελευταίο διάστημα. Και πολλοί από αυτούς που έχουν απολέσει αυτές τις θέσεις εργασίας δεν έχουν πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής ε, ασφάλισης και προστασίας και διάφορες ενισχύσεις που δίνονται από κυβερνήσεις σχετικά με την πανδημία. Επίσης δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή ε, ε, βασικά αγαθά όπως κατοικία, καθαρό νερό, δηλαδή στα πλαίσια της υγιεινής και της ε, αντιμετώπισης του ιού, της πανδημίας, αυτό είναι ιδιαίτερα πρόβλημα, είναι ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα και πώς μπορεί κανείς να ένα μαθητής να παρακολουθεί εξ αποστάσεω μαθήματα εφόσον δεν έχει σύνδεση ίντερνετ και δεν έχει υπολογιστή. Ε, και πώς θα λάβει το γεύμα που λαμβάνει από το σχολείο εφόσον κάθεται στο σπίτι και στηρίζεται σε αυτό. Είναι σημαντικό επίσης για τους Ρωμά να κάνουμε μία ανάλυση φύλου, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε βρει ότι οι εμπειρίες των Ρωμά γυναικών είναι πολύ δυσμενέστερες από εκείνες των ανδρών πάω στους ανθρώπους με αναπηρίες και στους πιο ηλικιωμένου. Και εδώ έχουμε ανησυχητικές τάσεις, μερικές από τις οποίες ήδη αναφέρατε. Έχουμε τον κίνδυνο σε κάποια ιατρικά κέντρα ε, κάποιου, αν θέλετε, κάποιας διαφορετικής αντιμετώπισης ή φιλτραρίσματος από πλευράς των υπευθύνων, όπου δεν τους κάνουν δεκτούς για εισαγωγή σε κέντρα πολλούς ηλικιωμένους δηλαδή, έχουμε διακοπή κοινωνικών υπηρεσιών και φροντίδας στο σπίτι, ιδιαίτερα για ανθρώπους με αναπηρίες, το οποίο έχει οδηγήσει σε πολύ συγκεκριμένα δεινά και δυσκολίες για τους ανθρώπους αυτούς. Επίσης ανισχυτικό στοιχείο είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε σε οίκους ε, αναπηρίας και τρίτης ηλικίας με άκαμπτα πλαίσια διοικητικά αν θέλετε τα οποία έχουν οδηγήσει σε ακόμα πιο αρνητικό αντίκτυπο για πολλούς ανθρώπους. Και έχουμε και το φαινόμενο που σε κάποιες χώρες ονομάζουμε κοκούνινγκ για τους ανθρώπους με αναπηρίες και τους ηλικιωμένους όπου δεν γίνονται σεβαστές οι εμπειρίες και οι επιδημίες των ανθρώπων αυτών δηλαδή. Όπως και στο χώρο εργασίας έχουμε ιδιαίτερα μειονεκτήματα και ε, έλλειψη επαρκούς δυνατότητας να ληφθούν τα μέτρα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Τώρα να πω μία λέξη για το, για το θέμα της ψηφιοποίησης της ζωής μας που προχωρεί ταχαίως αλλά έχει προκύψει ως ουσιαστικότατο ζήτημα στα πλαίσια των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στα πλαίσια της πανδημίας του COVID. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των προβλημάτων των ανθρώπων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων, η ψηφιοποίηση έχει οδηγήσει σε πολύ συγκεκριμένα εκτήματα. Δηλαδή, ιατρική φροντίδα εξ, εξ αποστάσεως, όπως θα μπορούσε να το πει κανείς, το οποίο είναι επιτυχής προσπάθεια, τουλάχιστον σε κάποιες χώρες, σε κάποια μέρη. Επίσης έχουμε ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση. Πέρα από, τα πλεονεκτήματα αυτά όμως, έχουμε πολύ μεγάλη επιδείνωση των μειονεκτημάτων που σχετίζεται με την πρόσβαση στο ίντερνετ, και σχετίζεται και με την παιδεία που δίδεται στα παιδιά των Ρωμά. Γιατί εδώ χρειάζεται hardware, χρειάζεται εξοπλισμό και χρειάζεται και πρόσβαση σε ένα επαρκέ σήμα. Ε, δηλαδή επαρκώς ισχυρό ίντερνετ αν θέλετε το οποίο είναι πολύ διαφοροποιημένο στις διάφορες χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωση και στις διάφορες περιφέρειες του. Υπάρχει το θέμα του ψηφιακού αλφαβητισμού όπου εκεί έχουμε πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ του πληθυσμού και μέρος των προκλήσεων στα πλαίσια του COVID για τις τρεις ομάδες που μιλούμε σήμερα και για αυτές είναι ο κίνδυνος διακρίσεων στην τεχνητή μας νοημοσύνη διακρίσεων κατά δηλαδή της τρίτης ηλικίας για παράδειγμα προκαταλήψεων ή διακρίσεων κατά της τρίτης ηλικίας τώρα επιτρέψτε μου να πω το εξής ε, παραμένουμε στον πυρήνα, στην καρδιά της πορείας της κρίσης αυτής. Καθόλου δεν έχουμε δει φως στο τούνελ. Και χρειαζόμαστε μεγαλύτερη προσπάθεια και εστιασμένη υποστήριξη των τριών ομάδων πληθυσμού που ανέφερα. Και ένα παράδειγμα συγκεκριμένη δράση που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι κοινωνική πρόνοια για τους Ρωμά. Και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να απαλύνουμε, για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες τους. Σε ευρύτερο πεδίο θα αναφερόμουν σε τρία στοιχεία που χρειάζονται την προσοχή μας. Καταρχά ο πυλώνας ε, των κοινωνικών δικαιωμάτων. Πρέπει να εμβαθύνουμε τα παραδοτέα, να βελτιώσουμε δηλαδή τα παραδοτέα του πυλώνα και στα πλαίσια του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την υλοποίησή του και αν θα μπορούσα να κάνω σήμερα εδώ μια έκκληση είναι να κάνουμε κάθε προσπάθεια που μπορούμε να εγγράψουμε τον πυλώνα σε συγκεκριμένα δικαιώματα. Έχουμε δικαιώματα που εγγράφονται στη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε μέσα του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά ίσως δεν εγγράφονται επαρκώς ε, οι πρακτικές, οι απτές διαδικασίες που οδηγούν σε αυτά τα δικαιώματα ή στην υλοποίησή τους. Και αυτό θα είχε σημαντική διαφορά. Δηλαδή, οι προϋποθέσεις για πλαίσια που να είναι διαφανή και πλαίσια λογοδοσίας σαφή θα ήταν σαφέστερη. Θα πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε τις προσαρμογές και αρκετά ταχαίως που χρειάζεται και όχι να μιλούμε απλώς για δικαιώματα των Ρωμά ή των λυκειωμένων ή των ανθρώπων με αναπηρία, αλλά τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες αυτές. Το άλλο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω σύντομα είναι ότι χρειαζόμαστε μια εξέταση του στρατηγικού πλαισίου που ανέφερε και η Επίτροπος. Είναι μια νέα ευκαιρία που πρέπει να την αρπάξουμε και θα πρέπει να φροντίσουμε τα παραδοτέα σε κάθε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε χωριό. Και τέλος, το τρίτο στοιχείο που ήθελα να αναφέρω είναι η επερχόμενη ενωσιακή στρατηγική για τις αναπηρίες. Θα ενθάρρυνα την Επιτροπή να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε η στρατηγική αυτή να αποτυπώνει πιστά τις δεσμεύσεις υπό τη συνθήκη που έχουμε συμμορφούμενοι προς τις ε, συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών για τις αναπηρίες. Θύμισα νωρίτερα ότι η προσέγγιση επί τη βάση των δικαιωμάτων βελτιώνει τα παραδοτέα. Και αγαπητά μέλη θα ήθελα να σας βεβαιώσω όπως πάντα για τη συνεχισόμενη δέσμευσή μας ως οργανισμό. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να εργαζόμαστε και να ενημερώνουμε την κοινωνία, να συντάσσουμε δελτία με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε απολύτω για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Μαζί με τα δεδομένα αυτά θα συνεχίσουμε και την έρευνά μας όπως για τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης επί των πληθυσμών τους οποίους εκπροσωπείτε και για την ανάπτυξη δυναμικού σε όλα τα κράτη-μέλη σε επίπεδο hardware και μέσων. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για τις τεχνικές δυσκολίες. found... Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φλάχερτη. Τα πορίσματά σας ε, τα έχουμε λάβει μέσω email και γνωρίζουμε πολύ καλά αναλυτικά το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής. Οπότε τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στον πρώτο γύρο ερωταπαντήσεων. Καταρχάς ε, θα ακούσουμε το Ελκα, την κυρία Ρώσα Εσταράς Φεραγκούτ. Δύο λεπτά θα έχει ο καθομιλητή στη διάθεσή του. Ε, Η κυρία Φεραγκούτ να πατήσει το κουπί speak. Γεια σας. Μ' ακούτε? Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε όπως και τον κύριο Φλάχερτη και την Επίτροπο. Διότι αυτή τη στιγμή πολλά είναι αυτά τα οποία μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν. Σίγουρα η πανδημία, μεγαλύτερος κοινωνικός αποκλεισμός, απομόνωση και σίγουρα αρνητικές επιπτώσεις για την αναπηρία και την ψυχική υγεία. Δεν έχουμε πλέον ε, την καθημερινή ρουτίνα τα άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένοι πλέον ε, έχουν γίνει ακόμη πιο ευάλωτοι. Πολλά τα προβλήματα για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας σε πολλά κράτη-μέλη. Υπάρχει επίσης πρόβλημα πρόσβασης, πληροφορίες, επικοινωνίας που επιδεινώνει την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε τώρα που είμαστε σε αυτή την κατάσταση πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις δυσκολίες την απομόνωση, τις δυσκολίες πρόσβασης. Επίσης, ε, όταν βρίσκονται σε κάποιο ίδρυμα αυτά τα άτομα, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα και με τους ηλικιωμένους και με τα άτομα με αναπηρία. Μεγαλύτερη απομόνωση, πολύ επιβλαβής. Και οι φροντιστές είχαν προβλήματα. Και για αυτούς είχαμε διαφορετική ρουτίνα. Επίσης, ενδοκογενειακή βία λόγω της απομόνωσης. Πρέπει λοιπόν να βρούμε δείκτες για όλα αυτά. Το σχέδιο ανάκτησης στο μέλλον, ανάκαμψη, συγγνώμη, θα πρέπει να βοηθήσει για τις ομάδες αυτές, ιδίω να είναι ένα σχέδιο ανάκαμψης αυτό που θα μπορέσει να διορθώσει τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει σε αυτή την περίοδο. Οι στρατηγικές για τα άτομα με αναπηρία σίγουρα θα πρέπει να αντλούν διδάγματα από την πανδημία. Το λέμε και στο ψήφισμά μας του Ιωνίου. Η στρατηγική αυτή πρέπει να λάβει υπόψη σε όλα αυτά. Την ψηφιοποίηση πρέπει να τη δούμε ως ευκαιρία. Μελέτη αντικτύπου ψηφιοποίησης. Πρέπει να δούμε όχι τις δικές μας ζωές πώς επηρέασε, αλλά και τα άτομα αυτά ιδιαίτερα, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. πρόσβαση υπηρεσίες, στις υπηρεσίες υγείας πρέπει να βελτιωθεί για τις αυπαθείς ομάδες. Αυτή η απαγόρευση ε, περιορισμός μετακινήσεων δεν θα πρέπει να συνεπάγεται απομόνωση. Ευχαριστώ. This Περάσατε βέβαια τα τρία λεπτά, λέει η Πρόεδρος. Θα παρακαλέσω όλους όσοι θα πάρετε το συνέχεια να μην υπερβούν το λόγο. Από τους σοσιαλιστές ο κύριος Μπέργλες. Δύο λεπτά παρακαλώ, το πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Ευχαριστώ τον κύριο Φλάχερτη και την Επιτροπή. Σίγουρα ο Οργανισμό των Δικαιωμάτων έχει να δραματίσει μεγάλο ρόλο. Πρέπει να δούμε πώ η πανδημία τη COVID-19 επηρεάζει αυτέ τι ομάδε για τι οποίε συζητούμε. αυτέ τι τρει ομάδε που μπήκαν ακόμα πιο πολύ στο περιθώριο, στο οποίο ήδη ήταν και πριν την πανδημία. Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν και επηρέασαν ε, τις ε, κατηγορίες αυτές του πληθυσμού περισσότερο από τις άλλες και αυτό μας ανησυχεί. Διότι στις μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν τα περισσότερα θύματα και, τα περισσότερα κρούσματα. Είμαι συγητής για τις εθνικές στρατηγικές για την εντάξει των Ρωμά και βλέπω πως οι Ρωμά και οι νομάδες αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Έχουν περιορισμένη πρόσβαση, παραδείγματος χάρη σε πόσιμο νερό. Η φτώχεια είναι οξυμένη. Υπάρχει λιγότερη κοινωνική προστασία. Η πρόσβασή τους ε, στο διαδίκτυο είναι ε, αποσπασματική. Αυτό επηρεάζει και τους νέους στην ηλικία ε, Ρώμα. Και βέβαια έχουμε και περισσότερες μολύνσεις από τον ιό του κορονοϊού μεταξύ των νόμων. Και αυτό οδηγεί σε έξαρση των προκαταλήψεων σε βάρος των τσιγκάνων θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί εδώ μιλάμε για πολλαπλές διακρίσεις. Είμαστε μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό γνωρίζει ότι θα ερχόταν αυτό το δεύτερο κύμα. Σας ερωτώ, είδατε κάποια βελτίωση στο ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των τριών αυτών ομάδων και στο πρώτο κύμα είδατε μήπως κάποιες καλές πρακτικές ό,τι αφορά την ένταξη των Ρωμά. Ποια είναι τα σημαντικά μέτρα εδώ. Ευχαριστώ. Πισλάρου Ρινιού, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Αγαπητή Πρόεδρε, αγαπητό τον κύριο Φλάχερτη και την Επιτροπή Ντάλη. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Δεν είχαμε προετοιμαστεί για αυτή την πανδημία σίγουρα, το ξέρουμε αυτό. Όμως περισσότεροι βασιζόμαστε στα προγράμματα κοινωνικής ε, πρόνοιας. Η Ρωμά όμως ε, είναι στα περιθώρια, είναι άσχημα συνθήκε διαβίωσης. Είναι μια συλλογική μας αποτυχία σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό. Δεν υπάρχουν σχέδια για αυτούς τους ανθρώπους. Ουσιαστικά θεωρείται και υπεύθυνοι γιατί ε, μεταδίδουν υποτίθεται την ε, πανδημία. Ε, στιγματίστηκαν οι Ρωμά. Απαράδεκτο αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, την ανάγκη για κοινωνική πρόσβαση, πρόσβαση στην υγεία και να μην παραγνωρίζονται τα δικαιώματα των Ρωμά, κάτι το οποίο έχει επιδεινωθεί. Όταν οι εθνικέ κυβερνήσει σε λίγο χρόνο και λίγη ε, δυνατότητα έχουν να αντιμετωπίσουν ε, όλα αυτά τα ζητήματα λόγω του αυξανόμενου αριθμού των κρουσμάτων. Τι έχετε να πείτε, τι μπορεί να κάνω στο πλαίσιο της δίκας λήψεως αποφάσεων για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σε επίπεδο στρατηγικής, σε επίπεδο κομισιών γίνονται πράγματα. Ποιε είναι οι προσδοκίε, τι δράσει μπορούν να ληφθούν, ο ρόλο του Κοινοβουλίου ποιο είναι για την αντιμετώπιση κατάσταση και σε ό,τι αφορά ε, και το άτομα με αναπηρία και του ηλικιωμένου που είδαμε φιαλτικέ σκηνέ την άνοιξη. Τώρα έχουμε το δεύτερο κύμα τι λύσεις εφαρμόστηκαν, τι λύσεις πρέπει να εφαρμοστούν για να προστατευτούν καλύτερα τα άτομα με αναπηρία απέναντι σε αυτή την πανδημία. Οι καλές πρακτικές που θεωρείται ότι πρέπει να προωθηθούν ποιε είναι και πώς μπορούμε να τις ε, μεταφέρουμε στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπίλτ για την ομάδα ID. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εδώ και κάποιου μήνε. Ε, Όλοι εδώ που μιλούν στηρίζονται και βασίζονται σε αυτή την υγειονομική κρίση και επαναλαμβάνουμε κάθε φορά αυτά που ξέρουμε πολύ καλά. Ενώ δεν ξέρουμε όμως με βεβαιότητα ο κόσμος αύριο πώς θα μοιάζει. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επωφελείται από την κρίση αυτή για να προωθήσει μια τζέντα. σήμερα συζητούμε για τους ηλικιωμένους, για τα άτομα με αναπηρία και ακόμη και για τους Ρωμά. Ας βάλουμε και τους μετανάστες μέσα, γιατί το κάνουμε σε άλλες περιπτώσεις. Τι σχέση έχουν όλα αυτά. Έχουμε μια σκανδαλώδη τακτική. Όλα αυτά που σπαθάμε στα επιβάλλεται ομού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μας κάνει κηρύγματα εδώ πέρα. Μιλά για τις ευπαθείς ομάδες. Ε, είναι πολύ του σειρμού αυτή η ορολογία και ουσιαστικά επιβάλλει στου Ευρωπαϊκού λαού πραγματικότητες που δεν τι θέλουν. Εγώ αυτό τον εκβιασμό δεν τον δέχομαι. Δεν θέλω με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίζουμε του Γάλλους που όλη τους τη ζωή έχουν εργαστεί και που πλήττονται ε, κατά μέτωπον από αυτή την κρίση και να του βάζουμε στο ίδιο καλάθι με του ε, τούντε άστελο, άσυλο ή μετανάστε που δεν έχουν δικαίωμα να είναι στη Γαλλική επικράτεια ή τα άτομα με αναπηρία που χρειάζονται ειδική βοήθεια δεν μπορούμε να του. Ε, ε, βάζουμε στο ίδιο καλάθι με τους χιλιάδες Ρωμά που δεν έχουν καμία δουλειά στη Γαλλία. Έχουμε ε, πολλούς από αυτούς να έρχονται από τη Ρουμανία. Είναι μέλος της Ένωσης. Δεν είναι πολιτικοί πρόσφυγες που διώκονται και υπάρχουν άστεγοι. Πάρα πολλοί άστεγοι. 300.000 στη Γαλλία, λέει ε, το Ίδρυμα Μπεπιέρ ότι είναι στη Γαλλία. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Συμφωνούμε όλοι ότι οι επιπτώσεις της κρίσης είναι φρικτές. Αλλά αφήστε μας το δικαίωμα να δούμε τους δικούς μας πρώτα και μετά τους άλλους. Ε, αυτό είναι ένα δικαίωμα, τουλάχιστον για μας τους Γάλλους. Ευχαριστώ πολύ. Ρωμαίο Φράντς τώρα, από τους Πράσινους. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Και θα ευχαριστήσω και τον κύριο Φλάχαρτη και την κυρία Ντάλη για τη δική του παρουσία. Το Σεπτέμβριο με 575 ψήφους υπέρ ένα ψήφισμα όπου αναφέρθηκε ακριβώς η κατάσταση που περιγράφεται και ε, συζητείται σήμερα για την Ευρώπη και το πώς κλειτάται από την πανδημία COVID-19, ιδίως ό,τι αφορά ε, Ρωμά. Συγκεκριμένα όμως πρέπει να τα πούμε τα πράγματα, η κατάσταση που βιώνουν οι περιθροπημένες ομάδες, η ε, Ρωμά μεταξύ αυτών, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι μια κατάσταση που την βλέπουμε, εγώ θα έλεγα εκατοντά, ε, ε, εδώ και δεκαετίες. Είναι αυτός, αυτή η προκατάληψη και ρατσισμός σε βάση των ε, τσιγκάνων είναι μια πολύ βαθιά και παλιά μορφή ρατσισμού και διακριτικής μεταχείρισης. Και δεν αναγνωρίζεται ότι υπάρχει στα εθνικά κράτη, ούτε και αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα. Χαίρομαι πολύ που με αυτό το ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που όπω είπα έγινε δεκτό με στριπτική πλησφιά, το αναγνωρίζουμε αυτό το πρόβλημα του ρατσισμού σε βάρο των τσιγκάνων. Και συνεργάζομαι πολύ καλά με την κυρία Νταλή. Αλλά αν θέλουμε να βελτιωθεί αυτή η συνεργασία, το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να το λύσουμε ρεαλιστικά. Πρέπει να υπάρξει δεσμευτικό χαρακτήρα θα πρέπει να υποχρεούνται τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τη δεκτική μεταχείριση και την, τον αριθμό σε βάρος των τσιγκάνων. Δεν το κάνουν αυτό μέχρι τώρα. Και θα πρέπει σίγουρα να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση ε, στην ε, ανάλυση και στην έβρεση λύσεων. Δεν θέλουμε πατερναλισμό, γιατί αυτό βγήκε και σε έλλειψη βιωσιμότητας και αηφορία στις λύσεις. Ε, όλα αυτά τα πράγματα τώρα συμβαίνουν και τώρα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το 2021 πρέπει να έχουμε μια νομοθεσία για την ισότητα, για την ισότητα μεταχείριση, ώστε αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα. και όλη η κοινωνία πρέπει να συμμετέχει. Να πω και κάτι στην προλαλή σας. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τις απόψεις και την προσέγγιση που έχετε εσείς. Όλοι είμαστε Ευρωπαίοι και όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Διακόπτεται. Sorry, you had your time. Sorry, this is almost three minutes. Okay, now the floor goes. Και τώρα. Κοιτάξτε, να σας πω ότι για χρόνια μας απασχολεί το θέμα για αυτούς τους ανθρώπους το ότι υπάρχει περιθωριοποίηση σε τόσα κράτη, υπάρχουν ε, δεσμενείς διακρίσεις και έχουμε ένα σωρό στρατηγικές, έχουμε περάσει ψηφίσματα για τους Ρωμά, αλλά δεν άλλαξε η κατάσταση. Άρα τα παχιά λόγια μέσα στα κείμενα αυτών των στρατηγικών δεν ωφελούν. Θα πρέπει να δούμε πώς τα κράτη-μέλη πρόκειται να έχουν στρατηγικές που θα βοηθήσουν αυτούς τους ευάλωτους ανθρώπους, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Και τώρα βλέπουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχει χειροτερέψει η κατάσταση κατά την πανδημία. Κύριε Φλάχερτη, πώς θα έχουμε το θαύμα, πώς θα κάνουμε τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να παίρνουν το θέμα αρκετά σοβαρά και να καταρτήσουν κάποιες πολιτικές που να τις εφαρμόσουν. Οπότε έτσι να βοηθήσουμε τελικά αυτούς τους ευάλωτους ανθρώπους. Και αυτές οι πολιτικές εντάσσονται στις πολιτικές για το κράτος δικαίου. Γιατί είναι ισχυρή μια κοινωνία όταν είναι ισχυρή η πιο ευάλωτη αυτής της κοινωνίας. Και τώρα, αφού σας τα είπα, τώρα η κυρία Πάλοπ από την Ενωτική Αριστερά. Κυρία Πάλοπ, πατήστε το κουμπί του μικροφόνου. Speak. Μάλιστα, μάλιστα, τώρα σας εντάξει, λέει η κυρία Πάλοπ. Ευχαριστούμε πολύ για τα όσα ελέγχθησαν και νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε τους τελευταίους μήνες ότι η πανδημία δεν έχει δείξει όλο το ίδιο. Οπότε θα πρέπει εδώ να δούμε τι γίνεται για κάθε ομάδα και οι τσιγκάλοι αυτοί, οι ΡΟΜ δυσανάλογα ε, χτυπήθηκαν και ακριβώς ε, πάθαν πάρα πολλά όπως αφορά την απασχόληση ε, τελικά ε, βρέθηκαν με κάποιες δουλειές που ε, δεν ήταν παραδοσιακές μορφές απασχόλησης, ήταν προσωρινές, οπότε έχουν πρόβλημα. Πάρα πολλά παιδιά δεν μπόρεσαν επειδή δεν έχουν ίντερνετ να συμμετάσχουν στο σχολείο από απόσταση και βέβαια λόγω των συνθήκων τους είχαμε περισσότερα κρούσματα και ε, βασανίζονται ιδιαίτερα οι γυναίκες που ε, φροντίζουν πολλούς. Έχουμε τώρα επομένω αυτό το πνεύμα εναντίον των ε, τσιγκάνων. Έχουμε σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Σλοβακία. Αλλά θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε για τα δικαιώματα όλων αυτών. Και είπαμε ότι έχουμε μία δέσμη μέτρων επανόρθωσης στην Ουγγαρία θα πρέπει να προστατευτούν αυτές οι μειονότητες, να αντιμετωπιστεί η ξενο... ξενοφοβία, ο ρατσισμό και να υπάρξουν δημοκρατικέ ελευθερίε που να γίνονται σεβαστέ, τα δικαιώματά του στην υγεία. Είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν πέρα από αυτούς τους στόχους του νέου στρατηγικού πλαισίου για την συμμετοχή, την ισότητα, όλα αυτά που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι λέτε κύριε Οφλάχερδε για όλα αυτά. Τι γνώμη έχετε. Ή ο Πρόεδρος. Και τώρα να μας πει ο κύριος ο Φλάχερτη να απαντήσει, αν μπορεί, τις ερωτήσεις μας. Μόλις πέντε λεπτά έχετε για όλες αυτές τις ερωτήσεις, κύριο Φλάχερτη. Έχετε το λόγο. Εσάς ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, θα κάνω ό,τι μπορώ. Μια σειρά από βουλευτές που έβαλαν ερωτήσεις, οπότε θα τις ομαδοποιήσω αν δεν σας πειράζει για τις βελτιώσεις όσον αφορά το τι γίνεται κατά την πανδημία με τους Ρωμά. Το πρόβλημα παραμένει πάρα πολύ σοβαρό. Σίγουρα αντιλήσαμε κάποια μαθήματα από όλα τα κρατημέλη. Να, για παράδειγμα, κάναμε το πείραμα να έχουμε κάποιους ε, διαμεσολαβητές, κάποιους ενδιάμεσους ε, για τις ανάγκες ε, των Ρωμά και αυτοί να είναι οι σύνδεσμοί τους με τις υγειονομικές αρχές. Αυτό το πείραμα πέτυχε. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον θεσμό και μετά την πανδημία να συνεχίσουν αυτοί οι ενδιάμεσοι, αυτοί οι διαμεσολαβητές να βοηθούν. Επίσης, όσον αφορά με την παιδεία από απόσταση, κανείς δεν ήξερε το Μαρτίο τι να κάνει, αλλά και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο ε, τα κέντρα αποφάσεων σε κάθε κράτος μέλος άντλησαν συμπεράσματα, αυτό ήταν εντυπωσιακό, ήταν και το θέμα επίσης των σχολικών γευμάτων που ξεκίνησαν τότε, θα συνεχιστούν τώρα και α έχουν κλείσει τα σχολεία γιατί είναι σημαντικό και επίσης όσον αφορά τα θέματα φροντίδα των ανηλίκων ε, το θέμα είναι σημαντικό για τα παιδιά για τις γυναίκες που τα φροντίζουν και όπου υπήρξε υποστήριξή τους αυτό ήταν μεγάλη βοήθεια. Έχουν βελτιωθεί τα θέματα τα θεσμικά, τα υγειονομικά, υπάρχουν στρατηγικές, βιωτικές ε, τους ε, συνθήκες, σε πολλά μέρη έχουν βελτιωθεί. Τώρα, πριν δούμε ε, άλλη ομάδα ερωτήσεων. Να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες ο οργανισμός μας εντυπωσιάστηκε από την δέσμευση των συστημάτων των κρατών μελών για πολλά ζητήματα και όχι μόνο για αυτές τις τέσσερις ομάδες που σήμερα συζητούμε, αλλά και τα δικαστήρια ήταν σημαντικά, τα κοινοβούλια που ανέπτυξαν ε, ιδιαίτερη δραστηριότητα, αλλά και οι εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, άλλαξαν κατεύθυνση, άλλαξαν το δίκαιο, τον νόμο, ούτω ώστε τα πράγματα να γίνουν πιο ανθρώπινα. Επίση είχαμε ένα σωρό ζητήματα. Το πώς, όπω είπε πρόεδρο, θα φέρουμε το θαύμα. Οι στρατηγικές δηλαδή για τους Ρωμά. Όλα επειδή επιδέχονται βελτίωση και η νέα μας στρατηγική έχει λάβει υπόψη συμπεράσματα που αντλήθηκαν ε, από το παρελθόν, από παντού και έτσι να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε εμείς την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, την πράξη δηλαδή, τι μάθαμε, τι συμπεράσματα πήραμε. Πρώτα-πρώτα ότι θα πρέπει να δρούμε σε τοπικό επίπεδο ε, και να μην είναι σε εθνικό επίπεδο μόνο στρατηγική να λαμβάνουν υπόψη οι, οι ρυθμίες της κάθε πόλης, του κάθε χωριού. Αυτά τα βρήκαμε δουλεύοντα επί τόπου. Και τους Ρώμα. Ε, θα πετύχουμε μόνο εάν και οι ίδιοι οι Ρώμα αγκαλιάσουν αυτή τη στρατηγική. Αν όλα αυτά γίνουν και εις βάθος, τότε θα αποδώσουν. Επίσης, τρίτον, το βασικό εδώ πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημα των Ρωμά, είναι το πρόβλημα δικό μας. Οπότε οι προσπάθειες να βελτιωθεί η κατάσταση των Ρωμά είναι κάτι το οποίο θα φέρει αλλαγές βαθιές στην κοινωνία και δηλαδή για όλο τον κόσμο θα σημαίνει ότι έγινε δουλειά με τις δυσμενείς διακρίσεις και με τον ρατσισμό. Άρα αυτό φορά και εμάς τους ίδιους αυτή η υπόθεση. Τώρα το τελευταίο να σας το πω γενικά για την βοήθεια προς τους Ρωμά θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση εργοδοσία και από τα φυσικά πρόσωπα και από τις αρχές. Και δημοσιονομικά, όσον αφορά ας πούμε ε, την στέγαση, αλλά και να δούμε τι γίνεται και με τα εγκλήματα μίσους κατά τον Ρωμά. Απέχουμε πολύ ακόμη από το να γίνουν αυτά πραγματικότητα. Επίσης, κυρία Μπίλτ, δεν ξέρω αν συμφωνώ με αυτά που είπατε, γιατί κάνετε τη διάκριση μεταξύ πολιτών και άλλων. Μα και οι Ρωμά είναι πολίτες στην κοινωνία μας. Και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν εξαρτώνται από το χρώμα του διαβατηρίου. Εξαρτώνται από το ότι κάποιος είναι άνθρωπος και έχει ανάγκες. Μα γιατί ακριβώς δίνουμε μάχες για να προστατεύσουμε από τον COVID ε, τους παππούδες μας, τους γονείς μας που είναι στα γυροκομεία, αλλά το ίδιο αφορά και τους Ρωμά. Όλους πρέπει να τους προστατεύσουμε. Όλοι δικαιούνται τη βοήθειά μας. Ακριβώς από σεβασμό για τα δικαιώματά τους και για την ιδιότητά τους ως ανθρώπων. Ευχαριστώ κύριε Να πάμε τώρα στον επόμενο γύρο ερωταπαντήσεων, λέει η Πρόεδρος. Έχετε ένα λεπτό και μόνο ο κύριος Μάντες από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ελπίζω να με ακούτε καλά. Έχω μια ερώτηση για τον κύριο Βλάτη. Μας μίλησε για φτώχεια, ένδια, ε, μεταξύ των ηλικιωμένων. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε αυτό και να επανεντάξουμε τους ανθρώπους αυτούς στην κοινωνία. Και δεν μιλώ για ένα κείμενο με ωραία λόγια. Τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο σύντομος, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Φεράντη από το S&D. Παρακαλώ. το κομβείο σας αν θέλετε. Ναι, σας ευχαριστώ. Ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για τις πολύ καλές εκθέσεις ε, σχετικά με τον αντέκτυπο της πανδημίας. Μιλώντας για τους ηλικιωμένους ε, και τους ανθρώπους με αναπηρίες όπως και τους φροντιστές τους που αντιμετώπισαν μεγάλα προβλήματα στην πανδημία, η κατάσταση μέσα στα κέντρα φροντίδας των ηλικιωμένων ήταν, υπήρξε δραματική σε πάρα πολλέ χώρε. Έχουμε προτάσεις ως ε, σοσιαλιστές για τη βελτίωση τη κατάσταση αυτής, αλλά καθότι έχω ένα λεπτό μόνο, ε, θέλω να αναφερθώ επιγόντω για μια οδηγία πλαίσιο που να συνοδεύει, που να, να πλαισιώνει την φροντίδα και την ε, κλινική και την οικιακή, και χρειαζόμαστε εναλλακτικά προγράμματα που βασίζονται στις τοπικές κοινωνίες, στις τοπικές κοινότητες. Το αίτημά μου προς τον οργανισμό είναι να έχουμε στοιχεία δεδομένα σχετικά με τις χώρες ε, εκείνες που έχουν ενσωματωμένα συστήματα φροντίδας στο σύστημα τους για την ψυχική και υλική στήριξη που χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Και εκμεταλλευόμενοι την ε, παρουσία της Επιτρόπου Ντάλι και διακόπτεται η ομιλήτρια για λίγο. Ε, ήθελα να μιλήσω για την ε, ε ίση μεταχείριση των διαφόρων πολιτών ανεξαρτήτως του φίλου τους, ε, το, της ε, φιλεκτικής τους ιδιότητος και να, να υπογραμμίσω ξανά την πολύ μεγάλη σημασία των φροντιστών του συστήματος φροντίδας. Είναι ε, ε, Ένα από τους πιο σημαντικούς πυλώνε του συστήματος κοινωνικής προστασίας που έχουμε. Σας ευχαριστώ. Ε, σας παρακαλώ κύριο Ζόρντι ε, από το Ρινιού. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε την Επίτροπο, ευχαριστώ τον κύριο Φλάιτη. Η Χάρτα Θεμελιωδιών Δικαιωμάτων στο κεφάλαιο 25 αναφέρεται στα δικαιώματα των ηλικιωμένων για αξιοπρεπή ζωή και διαβίωση αλλά εντός του COVID διαπιστώνουμε, διαπιστώσαμε και συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε ότι οι ηλικιωμένοι μας έχουν υποστεί ε, μεταχείριση απολύτως απαράδεκτη, απολύτως ελληματική. Αυτό είναι μια εικόνα που ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καταστάσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι ηλικιωμένοι και νομίζω ότι πρέπει να πάμε πέρα από διακηρύξεις και εκθέσεις και να κατανοήσουμε ότι οι ηλικιωμένοι μας είναι ευάλωτη ομάδα και χρειάζεται ιδιαίτερα μέτρα για την υποστήριξη και τη φροντίδη τους. Όπως έχουμε χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, χρειαζόμαστε μία, αν θέλετε, χάρτα ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, της τρίτης ηλικία. που να μην επιτρέψουν ποτέ ξανά να υποσκάπτονται τα δικαιώματά τους ε, και η φροντίδα που δικαιούνται να έχουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Φράνς έχει το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομος, κύριε Φράνς. Έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ πρέπει να πω κάτι ευχάριστο, ότι υπάρχει το REFIT που αντιμετωπίζει ακριβώς αυτά τα προβλήματα και στη Γερμανία και σε ε, άλλα μέρη έχει εφαρμοστεί ε, και το Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως και είπε ότι θέλει να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Η Κομισιόν θα πρέπει να έχει το σθένος να το εφαρμόσει αυτό, να τολμήσει να το κάνει. Και αν το κάνουμε είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση από κοινού. Έχουμε παραδείγματα καλών, βέλτιστων πρακτικών που λειτουργούν πολύ καλά εδώ και χρόνια και μπορούμε να τα εφαρμόσουμε σε όλη την Ευρώπη και δεν αφορά μόνο τα άτομα από την κοινότητα Ρωμά, αλλά και άλλε, τι περισσότερε σταθεροποιημένε ομάδε, άτομα με αναπηρία κτλ. Και θα βελτιωθεί η κατάσταση. Θα ήθελα να έχετε την τόλμη από κοινού με το Κοινοβούλιο να εφαρμόσει η Κομισιόν αυτά τα μέτρα. Για την ΚΟΥΕ τώρα έχει το λόγο η κυρία Πάλοπ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ε, όλοι έχουμε κατανοήσει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι μας σε όλες τις περιφέρειές μας, αλλά μας λείπουν δεδομένα, μας λείπουν στοιχεία, είναι κατακαιρματισμένη η εικόνα που έχουμε. Και θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Φλάιτη να μας δώσει περισσότερα δεδομένα για τις ε, λιγότερο καλές πρακτικές. Ε, στην Ισπανία είχαμε πολύ σημαντικό αντίκτυπο λόγω της ιδιωτικοποίησης πάραν πολλών φορέων ε, στα πλαίσια της υγείας και της φροντίδας. 22.300 και άνω ηλικιωμένοι σε, σε κέντρα τρίτης ηλικίας σε γυροκομεία και άλλα κέντρα έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία. Και επομένω, πρέπει να προσθεθεί και αυτό στο συνολικό κόστος ε, που έχει η πανδημία. Τι θα κάνουμε ώστε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα αυτά, τι θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε, να αναχαιτήσουμε την πρόοδο των ιδιωτικοποίησεων που οδηγεί σε αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Τελευταίος ομιλητής, η κυρία Γκέμα. Ένα λεπτό. Τζέμμα. Η κυρία Τζέμμα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Φλάιτσι. Δεν θα... Εννοείται ότι οι 200 και άνω εκατομμύρια άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολύ σημαντική ομάδα πληθυσμού. έχουμε αφήσει χωρίς καμία φροντίδα ευάλωτες ομάδες, πολύ ευάλωτες στο να, στην, ε, στο να προσληφθούν από τον ιό. Ο οργανισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων με τις εκθέσεις που έχει υποβάλει τις λεπτομερέστατες και που συμπεριλαμβάνουν πολλά στοιχεία, έχει καταγράψει αποκλήσεις, ε, μη συμμόρφωση προς τις, ε, τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται στα πλαίσια ε, γυροκομείων, κέντρων φροντίδας αλλά και φροντίδας οικιακής. Και ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε κάποιες οικονομικές λογικές και στρατηγικές προσεγγίσεις που έχουν χρεοκοπήσει ιδιαίτερα στα πλαίσια μιας τόσο σημαντικής πανδημίας και κρίσης. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε και πάλι τον κύριο Φλάιτι για πέντε λεπτά και μετά την Επίτροπο Ντάλι για άλλα πέντε λεπτά. Ο κύριος Φλάιτι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ε, βουλευτές. Υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με τους ηλικιωμένους. Θα εστιάσω σε αυτές καταρχάς. κύριος Μάντερς είπε πώς θα εντάξουμε κοινό στην κοινωνία τους ηλικιωμένους. Δύο απαντήσεις. Πρώτον, δεν θα πρέπει να τους στοχοποιήσουμε ως ε, ένα πρόβλημα. Θέλουν να συμμετέχουν ε, στο διάλογο, στην εξαίρεση λύσεων ηλικιωμένοι. Και δεν ακούγεται η φωνή τους επαρκώς. και με το ΖΡΟΜΑ και για όλες τις κατηγορίες. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε εμείς λύσεις για αυτούς αφήνοντάς τους εκτός. Δεύτερον, πρέπει να αναγνωρίσουμε ε, τις ε, εμπειρίες που έχουν ηλικιωμένοι. Δεν είναι μόνο η υγεία ή ε, το, η εμπειρία, η ηλικία τους. Είναι και το λεγόμενο διατομεακό στοιχείο και σε ό,τι αφορά το φύλλο. Οι ηλικιωμένε γυναίκε ε, αντιμετωπίζουν περισσότερε δυσκολίε από του ηλικιωμένου άντρε. Παραδείγματο χάρη, φρικτέ οι διαφορέ στη σύνταξη μεταξύ των δύο φύλων. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και το τελευταίο που έχω να πω για το πώ μπορούμε να στηρίξουμε του ηλικιωμένου στην κοινωνία είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε την ιδρυματοποίηση όταν αυτή η δύο είναι αχρίαστη. Μπορεί να απαιτείται κάποιες φορές και το δέχομαι. Πολύ κακή η σύνδεση του κύριο Φλάχερτη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φραντς που μας έδωσε το καλό παράδειγμα του Ρέφιτ στη Γερμανία. Θα το δούμε για την κυρία Ροτρίκες Πάλου μίλησα για το πρόβλημα δεδομένων. Εμείς συλλέγουμε υλικό για το 2020. Είναι και στα δημόσια δελτία μας αυτά τα στοιχεία. Τα έχω ανεβάσει στην πλατφόρμα σας. Αλλά έχουμε και στοιχεία αναχώρα, γιατί είπατε για την Ισπανία. Εκεί μπορείτε να δείτε σε κάθε μας, σε κάθε bulletin, στοιχεία πολύ λεπτομεριακά για την Ισπανία, τα οποία έχουν συλλέξει ερευνητικέ μας ομάδες. Πολλές πληροφορίες για πολλά θέματα ε, και σε σχέση με τους ηλικιωμένου. Στην πανδημία. Μιλήσατε για τις ιδιωτικοποίησεις και πώς επηρεάζουν, ιδίως τα δικαιώματα των ηλικιωμένων. Δεν θα τοποθετηθώ προς το αν είναι νόμι ή όχι ιδιωτικοποίηση ως πρακτική. Το θέμα είναι ότι ο ιδιωτικό τομέα, οι επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, να σέβονται, να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Νομίζω λίγο πολύ αυτά είχα να πω εγώ. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριο Φλάχερτη. Τώρα το λόγο έχει η Επίτροπος, κυρία Ντάλη, για πέντε λεπτά. Έχετε το λόγο. λεπτά. Πατήστε το κουμπί του μικροφόνου, λέει η γραμματεία στην κυρία Ντάλη. Can, can you hear me now? Ακούτε? Πολύ κακός ο ήχος, πάρα πολύ αντίχηση. Ευχαριστώ. Θα προσπαθώ να τα καλύψω τα θέματα που με αφορούν. Δεν ακούμε τι λέει η κυρία Ντάλη. Να μην αποδεπομπεί Ρωμά. Έχουμε το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου κατά τη ξενοφοβία του ρατσισμού και την οδηγία για την ισότητα των φύλων. Η Κομισιόν έχει ξεκινήσει διαδικασίε επί σε βάρο αρκετών κρατών μέλων. Ρωμά εντάσσονται και στο πλαίσιο της στρατηγικής κατά του ρατσισμού και εν μέσω πανδημίας έχω γράψει στους αρμόδους υπουργούς όλων των κρατών μελών και έχω τονίσει την ανάγκη να ληφθούν ειδικά μέτρα για τις ευάλωτες ομάδες, μεταξύ αυτών και για τους Ρωμά βέβαια, στο πλαίσιο της πανδημίας. Πρόσφατα είχαν το στρατηγικό πλαίσιο για την ισότητα της συμμετοχή για framework... Το πλαίσιο και η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που εγκρίθηκε από την Κομισιόν, όπως και το πλαίσιο, δίνουν κατευθυντήριες γραμμές. Θα βοηθήσει αυτά τα κράτη-μέλη να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν αντίστοιχε καταστάσεις στο μέλλον. σε ό,τι τη μελλοντική στρατηγική, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική στρατηγική, ξέρετε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις. Σημειώνω αυτό που είπατε για την ιδρυματοποίηση. Θέλουμε από ιδρυματοποίηση και το αναφέρουμε και στην στρατηγική. θέλουμε όλοι να συμμετέχουν στη δικασία αποφάσεων. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Στην στρατηγική, παραλαμβάνω, θα την υπόψη ο αντίκτυπος της πανδημίας και στο επόμενο θέμα της μερικής διάταξης θα σας αναφέρω πιο πολλά για αυτό το θέμα και τις συνιστώσεις. Τώρα, ηλικιωμένοι, εν καιρό πανδημίας, πήραν μέτρα τα κρατημέρια να μετριαστεί ο αντίκτυπος και αυτό επηρέασε και τα δικαιώματα και τη ζωή των ηλικιωμένων. Συστηματικές εξετάσεις, διαλογή στα νοσοκομεία, κοινωνική απομόνωση, πρόσβαση περιορισμένη στην υγειονομική περίθαλψη για τους ηλικιωμένους. Μεγάλη πρόκληση για τα κρατη που θέλουν να εξασφαλίσουν τη συνεχή πρόσβαση των ηλικιωμένων στις υπηρεσίε υγείας. Προσπάθουν και να συγκρατήσουν ε, την εξάπλωση της ε, νόσου. Είπατε πολύ και σωστά ότι έχει πληγεί περισσότερο αυτή η κατηγορία των ηλικιωμένων. Αλλάζει το δημογραφικό προφίλ. Έχουμε τη γύρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη που σημαίνει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολύ ομάδα, ιδίω αν λέμε υπόψη ότι και το 50% περίπου των ηλικιωμένων πάνω από 60 έχουν και κάποια μορφή αναπηρία. Άρα ακόμα χειρότερη κατάσταση. Πώ μπορούν να ζήσουν αυτόνομα, πώ μπορούν να ζήσουν εξωπρεπώ. Πολλοί ηλικιωμένοι ζουν μόνοι του. Μπορεί να μην έχουν εξοπλισμό ή να μην γνωρίζουν πώ μπορούν να εκμεταλλευτούν τα ψηφιακά εργαλεία για να δέχουν κάποιε επαφέ κοινωνικέ γιατί η απαγόρευση ή ο περιορισμός των φυσικών επαφών, σωματική επαφή έχει δημιουργήσει προβλήματα. Υπάρχουν περιοριστικά μέτρα σε πολλές χώρες και οι ηλικιωμένοι πλήττονται ακόμη περισσότερο. Άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι Ρώμα, άλλοι περιθωριοποιημένοι ε, πρέπει να υποστηριχθούν. Υπάρχει χρηματοδότηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή και της ε, οδηγίας, ε, μάλλον της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής για την αναπηρία. Εγώ σημειώνω τα σχόλιά σας ε, και θα τα λάβουμε υπόψη μας, θα τα λάβουμε υπόψη μας καθώς θα προετοιμάζουμε τη νέα στρατηγική την αναπηρία. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Ντάλη, λέει πρόεδρος. Ευχαριστούμε όμως και τους δυο σας, τους δύο προσκεκλημένους μας και νομίζω ότι τώρα με την ε, πανδημία θα έχουμε μια συνειδητοποίηση, ένα ξύπνημα πλευράς κρατών μελών για να προσέξουν τις πιο ευάλωτες ομάδες αναφέραμε, τους Ρωμά ε, τους ανθρώπους με αναπηρία αλλά και τους ηλικιωμένους. Όλα αυτά τα συζητήσαμε και ελπίζουμε ότι θα ληφθούν κάποια μέτρα τόσο ώστε αυτέ οι ευάλωτε ομάδε να υποστηριχθούν και επίσης ε, να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες φιλόδοξες στρατηγικές. Και συμφωνώ με τον κύριο Οφλάχερτη που μας εξήγησε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε, να προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων, αλλά θα πρέπει μαζί τους να προσπαθούμε να επεξεργαστούμε λύσεις Οπότε τώρα θεωρούμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η ανταλλαγή απόψεων και πάμε τώρα στο θέμα υπαριθμών 6. Πρόκειται για την ανταλλαγή απόψεων με την ε, Επίτροπο Έλενα Ντάλη για την ε, στρατηγική του το 2020 σε σχέση με τις ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί σε σχέση με το κείμενο, το σχέδιο γνώμη της κυρίας Λάγκεν ε, Ζήμπεν για το ε, ζήτημα το, του τι συνέχεια θα δοθεί ε, στο κείμενο το ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Τώρα, για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αναπηρίας μετά την περίοδο 2020, να μας μιλήσει η κυρία Ντάλη και κατόπιν η Κυρία Ντάλη, έχετε πρώτη εσείς το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Ντάλη. Και Η προηγούμενη στρατηγική από το 10 μέχρι το 20 ε, ακολουθήθηκε από κάποια αξιολόγηση ανεξάρτητη και μπορείτε να δείτε αυτή την τελική έκθεση μπορείτε να δείτε και μαζί και με το έγγραφο εργασία στο δικό μας όπου γίνεται κάποιος απολογισμός των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για την στρατηγική των ανθρώπων για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και τώρα οι συνεργάτες μας, οι υπηρεσίες μας επεξεργάζονται την ανακοίνωση της Επιτροπής για την μέλουσα ανακοίνωση για την περίοδο μέχρι το 30, από το 20 μέχρι το 30. Συνεργάζονται όλες οι υπηρεσίες της Κομισιόν με την αρμόδια γενική διεύθυνση. Λοιπόν, θα είναι πολύ άσχημος ο ήχος της κυρίας Ντάλη. Δεν ακούγεται καθαρά καθόλου. Οπότε, οι συναρμόδιες επιτροπές προσπαθούν, αλλά όλα αυτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα σε σχέση με τα προβλήματα για την αναπηρία. Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να δουν όλους τους σχετικούς τομείς και θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουν σε διαβούλευση γιατί θα γίνει ένας πρώτος γύρος διερευνητικός. Επίσης θα έχουμε μια δεύτερη σειρά συναντήσεων Οκτώβριο και Νοέμβριο. Ε, πρώτα ξεκίνησαμε το καλοκαίρι, ολοκληρώθηκε αυτός ε, ο άλλος γύρος Οκτωβρίου Νοεμβρίου, να δούμε όλα τα επιμέρους θέματα της στρατηγικής. Και κάνουμε τέσσερις θεματικές συναντήσεις για κινητικότητα, για συμμετοχή όσον αφορά την απασχόληση, τις δεξιότητες, κοινωνική πρόνοια, σχετικές υπηρεσίες και την ανεξάρτητη διαβίωσή τους, παιδεία, όλα τους τα δικαιώματα σε σχέση με την σύμβαση του ΟΗΕ και τα θέματα σχετικά με διακυβέρνηση όπως περιέχονται σε εκείνο το κείμενο ε, αυτού του οργάνου του ΟΗΕ. Έχουμε επομένω τώρα εισηγητέ από διάφορους κοινωνικούς φόρους, ε, πρόκειψαν διάφορα από αυτές τις τέσσερις συναντήσεις Οπότε έτσι γίνει μια καταγραφή τη κατάσταση ούτω ώστε να έχουμε την προπαρασκευή τη στρατηγική Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Κοινοβούλιο ε, έχουν, είναι στο ίδιο μήκο κύματο για το πώ θα πρέπει να προχωρήσουμε για να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Και όπω επανειλημμένα έχουμε πει για την στρατηγική που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον, θέλουμε να τα καλύψουμε όλα, όλα που καλύπτει το κείμενο αυτό, αυτή η σύμβαση του ΟΗΕ. Και θα θέλουμε να έχουμε μία προσέγγιση επί τη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίσης θα λάβουμε υπόψη το κείμενό σας στις 24 Σεπτεμβρίου για την εφαρμογή και υλοποίηση της οδηγίας 2078 78 Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το γενικό πλαίσιο όσον αφορά την ισότητα στην απασχόληση, ε, τη δουλειά ε, και η ευθυγράμμιση της ε, με τη σύμβαση του ΟΗΕ. Πολύ συχνά έχουμε αποστέρηση των δικαιωμάτων από αυτούς τους ανθρώπους όσον αφορά την απασχόληση. Δεν τηρούνται αυτά που λέει το άρθρο 15 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης και λέμε εμεί ότι θα πρέπει να έχουν αυξημένε αρμοδιότητε, οι αρχές ε, απασχόλησης θα πρέπει να υποστήριζονται αυτά τα πρόσωπα ούτως ώστε να μπορούν να μπουν και να κρατηθούν στην ε, αγορά απασχόλησης. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να βρουν κάποιους τρόπους. Θα πρέπει να γίνει προσαρμογή της κατάστασης και των ε, κρατικών υπηρεσιών ούτω ώστε η κατάσταση να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες αυτών των προσώπων. Να δούμε τι θα γίνει με την κατάρτισή τους ή τέλος πάντων τι δεξιότητέ του, ούτω ώστε να έχουν εξάρτητη διαβίωση, να μπορούν ενεργά να συμμετέχουν στα τη απασχόλησης και στην κοινωνία. Επίση, θέλουμε να υπάρχει αξιοπρεπής διαβίωση, στέγαση προσβασιμότητα στην ε, αγορά απασχόληση επίση. Οπότε διερευνούμε τι δράση μπορεί να αναλυφθεί όσον αφορά την παιδεία, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, ανάλογα με τι εθνικές αρμοδιότητες στον τομέα της ε, υγείας, γιατί υπεθεωρούμε ότι οι παρεμβάσεις για τη στήριξη αυτών των προσώπων στα πλαίσια ε, του να υπάρχει μία παιδεία χωρί αποκλεισμού, είναι κάτι που θα πρέπει να καλυφθεί από αυτή την στρατηγική. Και η δικαιοσύνη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, αλλά και όλες οι κοινωνικέ οργανώσεις. Δηλαδή, να υπάρχει αμοιβή αναγνώριση του καθεστώτος ε, των προϋποθέσεων για να χαρακτηριστεί κάποιος ε, ανάπηρος, να υπάρχει σχετική κάρτα παντού Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Ανεξάρτητη διαβίωση. Ε, αυτό να είναι ένας θεσμός. Αυτό να είναι κάτι το προβεβλημένο, αναγνωρισμένο. Θα πρέπει να μπορούν ε, αυτά τα πρόσωπα να διαλέξουν πού και με ποιον θα ζήσουν. Και επίσης οι δημοτικές υπηρεσίες ε, θεσμικά να βοηθούν με βάση τα κοινοτικά κονδύλια. Στοχευμένες να είναι οι υπηρεσίες, και έτσι να μην γίνεται αποκλεισμό αυτών των πρόσωπων, να συμμετέχουν παντού στην κοινωνία. Πληροφόρηση. Προσβάση. Και αυτό θα πρέπει να καλυφθεί. Επίσης να δούμε και τι γίνεται με το δικαίωμά τους στο να συμμετέχουν στο δημοσίο βίο, στον πολιτικό βίο, το εκλέγει, το εκλέγεστε το 2024 τις επόμενες εκλογές θα πρέπει όλα τα θεσμικά όργανα να προσπαθήσουν να υλοποιήσουν αυτόν τον στόχο. Θα πρέπει εμεί να είμαστε το παράδειγμα προς μίμηση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Να μπορούν να έχουν εκλογικά κέντρα που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα πρόσωπα αυτά. εμείς τι θα πρέπει να διευκολύνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Το περιβάλλον. Από πάσα απόψη θα πρέπει να είναι συμβατό, να είναι όλα προσβάσιμα. Θα πρέπει όλα αυτά τα αισθήματα να μπουν στην κοινωνική νομοθεσία, στι πολιτικέ, να γίνει mainstream και σε στενή συνεργασία και με τα άλλα θεσμικά όργανα. Και έτσι να έχουμε συντονισμό, Ούτως ώστε να ελοποιήσουμε τη σύμβαση του ΟΗΕ ε, και θα ληφθεί υπόψη όπως είπαμε το ψήφισμα του Ιουνίου. Επίσης, συμμόρφωση με όλα όσα προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναπηρία, παντού όπου υπάρχουν ε, ανθρωπιστικοί πόροι και συμμόρφωση, επομένως με τις διατάξεις του ΟΗΕ. Αυτό είναι στόχος μας για την επόμενη δεκαετία. Να αλλάξουν τα στερεότυπα. Να σταματήσει ο στιγματισμός. Πολύ σημαντικό. Έτσι θα θωρακίσουμε αυτά τα δικαιώματα. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να υπάρχει συνειδητοποίηση του θέματος σε όλα τα επίπεδα. Συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να μπορέσουμε η πρωτοβουλία αυτή να πετύχει. Ευχαριστούμε την κυρία Επίτροπο. Η κυρία Λάγκεν Ζήπα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Dear Chair, dear colleagues. Αγαπητοί πρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω θερμά και να καλωσορίσω την Επιτροπό, την κυρία Ντάλη, που είναι μαζί μας σήμερα για να μας ενημερώσει για το πώς έχουν τα πράγματα για την προετοιμασία της ε, στρατηγικής για τις αναπηρίες μετά το 20. Τον περασμένο Δεκέμβριο εκ μέρους των Πρασίνων είχα ζητήσει ένα ψήφισμα για τη στρατηγική μετά το 2020. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ε, στρατηγική για τις αναπηρίες και το επιθυμητό της περιεχόμενο. Ελπίζω ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που καθυστέρησε λόγω του κορονοϊού και υιοθετήθηκε μόνο τον Ιούνιο, να έχει αποσταλεί στο γραφείο σας, να το γνωρίζετε και ελπίζω τα αιτήματά μας να ληφθούν αρκούντος υπόψη σας ώστε να διαμορφώσετε σωστά τη στρατηγική αυτή για μετά το 2020. Αγαπητή κυρία Ντάλη, η πραγματικότητα είναι δυστυχώς ότι δεν σεβόμαστε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα ανθρώπων με αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Είναι δυστυχώς η πραγματικότητα ότι όλες οι αρχές και οι αξίες μας που αποτυπώνονται στις συνθήκες μας δεν σημαίνουν τίποτα για τους ανθρώπους αυτούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, διακρίσεις για την πρόσβαση στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, στη σεξουαλική τους υγεία, στο δικαίωμά τους να ζουν ανεξάρτητα και αξιοπρεπώς, στην πρόσβασή τους στις συγκοινωνίες, στις επικοινωνίες, και στην αντιμετώπιση φαινομένων βίας. Χιλιάδες συμπολιτών μας, χιλιάδες εξημών δηλαδή, είναι αναγκασμένοι να μένουν σε διαφορετικά κέντρα υπό διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης από αυτές που θα μπορούσαμε να έχουμε στο σπίτι μας Και όλα αυτά συμβαίνουν παρά την εργασία που κάνουν διάφορες διεθνώς μη καπαομικρόν και καταγράφουν τις ελλείψεις αυτές, τις αποκλήσεις αυτές, τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν πολλοί από εμά ξαναλέω. Και επομένως σχετικά με τη στρατηγική για μετά το 2020 Πιστεύω ακράδαντα ότι χρειαζόμαστε μια πληρέστατη και απολύτως φιλόδοξη στρατηγική. Πρέπει να αποφύγουμε μια επιλεκτική προσέγγιση και να πάμε σε μια πληρέστατη προσέγγιση με φιλόδοξους στόχους υλοποίηση, φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα που θα ενταχθούν στο πλαίσιο διακυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, μια στρατηγική που θα αντιμετωπίζει τι συγκεκριμένε προκλήσει και δυσκολίε των ανθρώπων με αναπηρίες που υφίστανται διατομεακές διακρίσεις. Και δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι με αναπηρίες απολύτως ομοιογενής ομάδα. Είμαστε άνδρες, γυναίκες, είμαστε διαφόρων προελεύσεων και εθνικοτήτων. Υπάρχουν διάφορες διακρίσεις που δεν μπορούν να διαφεύγουν της προσοχής μας. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική που να μπορεί να προσαρμοστεί στις διάφορες περιοχές πολιτικής υπό τις συνθήκες της κρίσης της πανδημίας του COVID. Χρειαζόμαστε εστιασμένα μέτρα δηλαδή, στοχευμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τις σοβαρότατες αυτές δυσκολίες και τις παραβιέσεις των θυμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρίες. Και η στρατηγική αυτή θα πρέπει να συνδιαμορφωθεί μαζί με τους ανθρώπους με αναπηρίες και τις οργανώσεις, τους φορείς που τους εκπροσωπούν. Αυτή η δουλειά θα πρέπει να γίνει από εσάς, από την Επιτροπή. Και θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν και το σύνολο των νομοθετικών διατάξεων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη προσοχή που θα πρέπει να δίδεται στην καταπολέμηση των φαινομένων βίας. Και ολοκληρώνω, Πρόεδρε, χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτική για τις αναπηρίες μετά το 2020 και επιγόντως χρειαζόμαστε την υιοθέτηση της ε, προτινόμενης οδηγίας για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, της οριζόντιας οδηγίας. Ευχαριστώ, ε, λέει η Πρόεδρος. Θα πάμε τώρα στον πρώτο γύρο ερωταπαντήσεων. Ο κάθε ένας από εσά θα έχει δύο λεπτά για τις ερωτήσεις σας. Ξεκινάμε το ΕΛΚ. Ο κύριος Κόσα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας μάλλον να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους σας για τις τοποθετήσεις να σχολιάσω καταρχάς το σχέδιο έκθεσης και τις τροπολογίες. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλή ενημέρωση για το κείμενο. Νομίζω ότι και οι τροπολογίες που ε, θα υποβληθούν είμαι σίγουρος ότι θα είναι εξαιρετικές. Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ μαζί σας επ' αυτού. Για τη νέα στρατηγική και τα όσα είπε η Επίτροπος, είναι πάρα πολύ σημαντικό η νέα αυτή στρατηγική όχι μόνο να συνοψίζει το τι συνέβη την περασμένη δεκαετία, αλλά να μας δίδει νέες κατευθύνσεις για το μέλλον. Συμφωνώ απολύτως με κάποια από τα σχόλια που ακούστηκαν. Πιστεύω ότι η επιτήρηση, η παρακολούθηση των μέτρων θα πρέπει να ενισχυθεί. Και τι εννοώ. Χρειαζόμαστε δημοσιονομικούς πόρους, χρειαζόμαστε πόρους και μάλιστα σημαντικούς πόρους προκειμένου να υλοποιηθεί η νέα στρατηγική μέχρι το 2030. Όπως και χρειαζόμαστε πόρους για την παρακολούθηση των μέτρων αυτών και υπάρχουν κάποιοι ορισμοί που θα πρέπει να διευκρινιστούν, να αποσαφινιστούν. Χρειαζόμαστε καθοδήγηση για την παροχή διαφορών υπηρεσιών πρόνοιας, υγείας, μεταφορών, ίσης ε, πρόσβασης στην αγορά στην εργασία μην ξεχνούμε ότι μπορούμε να έχουμε το καλύτερο νομοθέτημα αλλά αν δεν υλοποιηθεί δεν θα έχουμε καταφέρει τίποτα. Λόγω των οποίων τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υλοποιήσουν πλήρως τη νέα νομοθεσία. Η νέα στρατηγική είναι ένα καλό πλαίσιο μελλοντικής συνεργασίας και ελπίζω να είναι και φιλόδοξη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άγχελες Εντί, παρακαλώ. Δύο λεπτά. Αν θέλετε να, απαντήσετε, να πατήσετε το κομβίο. Ναι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Επιτρόπο. Αναφέρθηκε στην έκθεσή μας του Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την, ε, ε, ε την ε, εισηγήτρια την κυρία Λάγκεν Τζίπν είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε πολύ καλούς συμβιβασμού. Είναι τόσο εξαιρετική η βάση, η δουλειά που έχω γίνει, που δεν έχουμε και πολλή δουλειά μπροστά μας από αυτού. Ευχαριστούμε κάτρι. Τώρα, γνωρίζουμε ότι κάποια δεδομένα που έχουμε στη θέση μας δεν είναι και τόσο καλά. Δεν αποτυπώνουν δηλαδή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρίες, το διαφορικό μισθόν τις δυσκολίες μεταφοράς και πρόσβασης στον χώρο εργασίας, μεταξύ άλλων. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ισχυρότατη στρατηγική για τις αναπηρίες. Για τα δεδομένα ήθελα να πω ότι έχουμε σημαντικές ελλείψεις συλλογής δεδομένων, ιδιαίτερα για αυτούς που μένουν εκτός κατοικίας σε κέντρα υποδοχής, σε οποιοδήποτε φορέα φροντίδας. Ε, και τα, το πρωτόκολλο ε, στο CRPD είχαμε ζητήσει να ε, επικυρώσουμε και τη συνθήκη της Ίσταμπουλ ε, είχαμε ζητήσει καλύτερη υλοποίηση σε, σε επίπεδο προσβασιμότητας είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό για τη στρατηγική και επίσης έχουμε ζητήσει από το Συμβούλιο να ξεμπλοκάρει ξανά και ξανά έχουμε ζητήσει την οριζόντια οδηγία πλαίσιο κατά των διακρίσεων. Και έχω και κάποιες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, αν μπορώ. Το μελλοντικό θεματολόγιο για τις αναπηρίες, για την εξέβρεση εργασία από πλευρά των ανθρώπων με αναπηρίες, αλλά και την αντιμετώπιση της ένδυας παρά τη θέση απασχόλησης. Επίσης αναφέρθηκε η Επίτροπος ε, για την κάρτα και την ενίσχυσή της. Δηλαδή εννοεί ότι θα πάει πέρα από θέματα αναψυχής. Επίσης η Επιτροπή πώς θα αντιμετωπίσει τις δυσκολίες των ανθρώπων με αναπηρία όταν μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος. Θα προτείνετε δράσεις για να εξασφαλίσουμε ομοιόμορφη αντιμετώπιση των δυσκολίων αυτών στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Από το Ρινιού, κυρία Μάξοβα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε Τάλη, αγαπητοί συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια είδαμε πολλά νομοθετικά επιτεύγματα για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. συμμετέχουν μεν περισσότερο και οι ονόσεις αυτών των ατόμων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν βλέπουμε να λαμβάνεται υπόψη ακριβώς πραγματικότητα ε, σε ό,τι αυτά τα δικαιώματα αυτών των ατόμων. Για να βελτιωθεί η κατάσταση και να μειωθούν οι φραγμοί, τα εμπόδια, πρέπει να συλλέγονται δεδομένα. Αλλά αυτό αποτελεί πρόκληση, ιδίως στο πλαίσιο της μελλοντική στρατηγικής για την αναπηρία είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό το πρόβλημα. Επηρεάζεται και το μέσα απασχόλησης. Αν θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, όπου υπό εκπροσωπούνται αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να μπορούμε να μετρούμε την πρόοδο που επιτελείται Αυτό αφορά και την αγορά εργασία και την παιδεία και την εκπαίδευση, κατάρτιση. Επίσης, σε αυτή την περίοδο ε, που έχουμε επιτάχυνση της ψηφιοποίηση και οικολογική πράσινη μετάβαση, ακόμη περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ανάγκε των ατόμων με αναπηρία. Πράσινη συμφωνία θα δημιουργήσει δεκάδε χιλιάδε νέες θέσει εργασία. Πόσες από αυτέ θα ε, τις πάρουν ε, άτομα με αναπηρία, πόσα ε, άτομα με αναπηρία θα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση. Τελικά η ανάγκη είναι να ληφθεί υπόψη σε όλα τα νομοθετήματα η διάσταση της αναπηρίας. Γι' αυτό, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι διατάξεις και της σύμβασης του ΟΗΕ, γιατί μας δίνει μια ισχυρή εντολή και πρέπει να λάβετε όλα τα θεσμικά όργανα υπόψη τα άτομα να αναπηρία, στην στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάξοβα. Κυρία Ζαμέ τώρα, ID. Ευχαριστώ αυτοί συνάδελφοι. Είναι η χρονιά για την αναπηρία και πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζεται η αναπηρία στις κοινωνίες μας. Δυστυχώς, αν δει την καθημερινότητα με τον φακό μου στον παραμορφωτικό, ουσιαστικά δεν θα δούμε τις πραγματικές δυσκολίες ε, και ε, τα βάσανα που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν πολλά προβλήματα. Δεν το αρνείται κανείς. Πρόσβαση. Σημαντικό πρόβλημα η έλλειψη προσβασιμότητας ιδίω για τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει ε, να κάνουν ολόκληρο αγώνα για να μπουν σε ένα λεωφορείο ή ε, στα μέσα συγκοινωνία στα άλλα, να αλλάξουν πεζοδρόμιο, να ανέβουν ε, επίπεδο κτλ. Ε, ή η πλαισίωση. Στη Γαλλία έχουμε πολλά προβλήματα. 2,7 εκατομμύρια είναι αυτά τα άτομα. Πέφτουν σιγά σιγά τα στερεότυπα όμως έχουμε διπλάσια ανεργία σε αυτή την κατηγορία. Αν δει για ποιο λόγο κανεί όμω δεν προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία επιχειρήση, το πρώτο εμπόδιο είναι η εκπαίδευση. Άρα αυτό μας παραπέμπει στο πρόβλημα ότι δεν είναι αντιληπτή η σχέση μεταξύ ε, των πολιτικών επαγγελματική κατάρτισης και των αναγκών για δεξιότητες. Άρα πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη και μένει πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυστρία, Σουηδία. 60% των ατόμων με αναπηρία έχουν θέση απασχόληση, έχουν δουλειά. Πρέπει να φτάσουμε τι χώρε αυτέ και να τα δούμε τα θέματα χωρί ιδεολογικέ ε, περιορισμού, ιδεολογικούς περιορισμούς. Δεν πρέπει να περιμένουμε θα πούν οι Βρυξέλλες. Κύριο Φλάχερτ, η εθνική προσέγγιση δουλεύει χωρίς ε, ε ιδεολογίες βλαπτικές. Αυτό είχα να πω. Ευχαριστώ, ECR. Ντελαπίσα. Δεν ακούγεται. Uh, we can't hear you. Maybe your microphone is muted. Now, now we can hear you. Yes. Είχατε κλειστό το μικρόφωνο, μήπως; Σας ακούμε τώρα, σας ακούμε τώρα λέω. Χάθηκε η κυρία Ντελαπίσα όμως. Now. Τώρα με ακούτε. Με ακούτε πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Αγαπητή Επίτροπε, ανησυχεί για τα μαμενα πήρα η Κομισιόν πρέπει όμως να βοηθήσει πραγματικά και αυτό δεν το κάνει. Ε, μυρολατρικά τα βλέπουμε. Λάθος προσανατολισμός για τη στρατηγική. Στην Ισπανία υπάρχουν όμως ε, πολλά προγράμματα που τα μας κάνουν αισθάνομαι υπερήφανους. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για κάποιες καταχρήσεις, αν είναι συστηματικές αυτές οι καταχρήσεις και να θυματοποιούμε αυτούς τους υποτιθέμενε βάλου τους πολίτες τα άτομα με αναπηρία πρέπει ε, φυσιολογικά να συμμετέχουν στην κοινωνία, να θεωρείται κάτι φυσικό αυτό. Ελπίζουμε με ελπίδα να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Μας ανησυχεί ο τρόπος με τον οποίο τροποποιείται αυτή η οδηγία. Αντί να βελτιώνει, μπορεί να γίνει παγίδα. Προτείνει ενεργή, ε, ενεργό συμμετοχή στον εργασιακό βίο. Δεν λαμβάνει υπόψη ότι σαστικά μιλάμε για πολύ διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ομοιογενή αυτή η ομάδα. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου, να δίνουμε επιλογές. Πρόστιμα, κυρώσει. Δεν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση, γιατί δεν λύνουν το 10, που είναι το πιο επίμαχο. Μιλάμε για αυτά τα εργαστήρια ε, προστατευόμενα, αλλά δεν βλέπουμε ε, τις διαφορετικότητες, ε, τις ιδιαιτερότητες. Δεν θα πρέπει να επηρεαστούν από την οδηγία, παράδειγμα χάρη τα εργαστήρια εργασιακής θεραπείας ε, ή άλλα εργαστήρια. Μην τα συγχαίουμε όλα. Γιατί αυτά τα προστατευόμενα εργαστήρια που δίνουν ζωή σε άτομα με μεγάλες ανάγκες ε, θα τα παραλύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δελαπίσα, και έκλεισε επομένως αυτός ο πρώτος ε, γύρος ερωτήσεων, αλλά έχουμε και για αυτόν τον γύρο και την κυρία Περέιρα για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ε, κυρία Ντάλη που ήρθε να μας μιλήσει Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο της όσον αφορά του αναπήρους οι οποίοι δικαιούνται να έχουν μια ανεξάρτητη ζωή χωρίς περιορισμούς, να υπάρχει ε, στην πράξη προσβασιμότητα στις σχετικές ε, υπηρεσίες, να υπάρχουν επομένως τα περιθώρια για ε, μια ζωή με ποιότητα. Θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας όσον αφορά τα δικαιώματά τους, θα πρέπει με αξιοπρέπεια να μπορούν να καταρτίζονται ε, θα πρέπει να είναι συμβατά με τις ανάγκες τους και τα ωράρια εργασίας, συνθήκες εργασίας, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσιους χώρους, σε μεταφορές, στα κτίρια. Ε, οπότε θα πρέπει να γίνει σχετική επένδυση, ε, να υπάρχει μια τέτοια παιδεία, να υπάρχουν κάποια δίκτυα ε, της προσφοράς φροντίδας και υπηρεσιών και κατοίκων, οπότε θα πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία με όλους, όλους μας που ασχολούμεθα με αυτό το ζήτημα, να καλύψουμε επομένως ε, όλη την υστέρηση που έχουμε όσον αφορά το να δώσουμε μια συνέχεια στο κείμενο, στη σύμβαση ε, του ΟΗΕ, να δείξουμε στην πράξη την ελεγγύη μας και επίσης να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Τώρα, θα σας ρωτήσω, κύριε Επίτροπε, θέλει με συγκεκριμένες προτάσεις η Κομισιόν να προσχωρήσει, να χρηματοδοτήσει ε, του δημόσιες φορείς ούτως ώστε να μπορούν να προσφερθούν οι σχετικές υπηρεσίες και τελικά τα πρόσωπα αυτά να μπορούν να είναι οι ωφελημένοι. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει ο Πρόεδρος και τώρα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή Ντάλη για να απαντήσει. Έχετε πέντε λεπτά κυρία Ντάλη για να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Ms. Dali, press the speak button, please. Είστε το κουμπί του μικροφόνου σας, κυρία Ντάλη. Μάλιστα. να προσπαθήσω σε σχέση με το ψήφισμά σας. Έχει διόντως ληφθεί υπόψη στην προετοιμασία της στρατηγικής. Οπότε και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε την πορεία για την υλοποίηση της σύμβασης του ΟΗΕ. Βεβαίως και χρειαζόμαστε την πλήρη συνεργασία των κρατών μελών. Προς τούτο. Τώρα για το θέμα του οριζόντιου χαρακτήρα της στρατηγικής δεν είναι δυνατόν αλλιώ να έχουμε πλήρη στρατηγική χωρίς να ισχύει μια, ένα τέτοιο ένα, ένας τέτοιος χαρακτήρας που δηλαδή ότι θα πρέπει να διαπνεί όλους τους τομείς και επίσης ο, το κάθε πρόσωπο είναι διαφορετικό από το άλλο οπότε και τα πρόσωπα με αναπηρία δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα, όπως δεν υπάρχει καμία ομάδα προσώπων που να έχει ομοιογενή. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιου είδους ε, ε, στρατηγική που να διαπνέει κάθε τομέα. Για όλους, για, όλους όμως και για τους ε, θα πρέπει η στρατηγική μας ε, για τους ΛΟΑΔΓΙ να καλύπτει το, επίσης τους αναπήρους και για όλους, για όλους. Άρα να υπάρχει αυτός ο χαρακτήρας ότι διαπνέει στρατηγική κάθε τομέα, κάθε, κάθε ομάδα. Οι στρατηγικές αυτές να αποτελούν μία ε, ουσιαστικά και επίσης ε, ε, να καλύπτονται κατά αυτόν τον τρόπο η κάθε μία από αυτές τις ομάδες. Είτε μιλούμε για ισότητα φίλων, είτε μιλούμε για ΛΟΑΔΚΙ, και η ομάδα των πρόσωπων με αναπηρία. Όλοι, όλοι έχουν ε, ε, διαφορετικές ανάγκες. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει τέτοιο χαρακτήρας ε, οριζόντιος και εγκάρσιος. Είπαμε για ανεξάρτητη διαβίωση και είπαμε ότι θα πρέπει να μην υπάρχει ε, κάποιο είδου ε, ε, ιδρυματοποίηση και σε όλη την ε, μακρά διαβούλευση πάντοτε θέλαμε να μην υπάρχει τέτοια ιδρυματοποίηση. Πάντα πάντα αυτό ήταν μια σταθερή σε όλες μας τις επαφές και συζητήσεις. Επίσης, θέλουμε να βλέπουμε μπροστά με αυτή τη στρατηγική ορθώς ελέγχθη ότι αυτή η στρατηγική είναι τμήμα μόνο της όλης διαδρομής. Χρειάζεται να συνεργαστούν πλήρως τα κρατη Απασχόληση. Ακριβώς όπως ελέγχθη. Διακόπτεται η κυρία Ντάλη. Η σύνδεσή της διακόπηκε. Τα είπαμε στην αρχή για την απασχόληση. Θα πρέπει όπου υπάρχουν κενά να αρθούν. Μία αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Να αξιοποιήσουμε το δυναμικό, τις δυνατότητες, τα ταλέντα, τις δεξιότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με την παιδεία, με την ενθάρρυνση για ανεξάρτητη διαβίωση, Κόβεται πάλι η φωνή της κυρίας Ντέλ. I take note of your point and the gaps in... Έλαβα υπόψη αυτό το που είπατε, ότι υπάρχει πρόβλημα με τα δεδομένα και έλαβα υπόψη και με τα σχόλιά σας για επέκταση της ισχύω της κάρτας αναπηρίας. Να δούμε πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά, τι θα γίνει με τις υπηρεσίες φροντίδας. Μιλούμε για συγκεκριμένη εκπαίδευση των προσώπων που προσφέρουν τη φροντίδα. Αυτό θα πρέπει φυσικά να περιλαμβάνεται στη στρατηγική. Και επαναλαμβάνω ότι θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο θέμα των δικαιωμάτων ανθρώπων με αναπηρία. Είναι, είναι για μας κορυφαία προτεραιότητα. Βεβαίω θα πρέπει να υπάρχει φροντίδα τη διακίνησή τους, να αρθούν τα εμπόδια για να μπορούν να διακινούνται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μετακινούνται και το έχουμε και αυτό ως προτεραιότητα. Οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επεξεργαστεί την υπόθεση αυτή συντονισμένα. Γι' αυτό, γι' αυτό και έχουμε τι στρατηγικέ σαν αυτή που συζητούμε. Βασικός φραγμός στην ελεύθερη διακίνηση είναι ότι δεν υπάρχουν τα αναγκαία πλαίσια και φυσικά έχει να κάνει εδώ και το πρόβλημα των δυσμενών. Σα σας διακόπτω, σας διακόπτω κύριε Ντάλιλε πρώτος, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε τώρα λήξη της ε, πρώτης ψηφορίας. Και έχουμε τώρα τη δεύτερη ψηφοφορία η οποία θα γίνει αύριο. Αύριο στις 11.30 και θα κρατήσει μέχρι τις 12 και 4. Και τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε τον δεύτερο γύρο των ερωταπαντήσεων. Αλλά έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω για το χρονικό μας πλαίσιο. Οπότε θα σταματήσει η διερμηνία. Πρέπει να φύγουν οι διερμηνείς και οπότε θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τα αγγλικά. Όποιος δεν καταλαβαίνει τα αγγλικά θα έχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Δεύτερος γύρος όλα τα απαντήσουμε. Ο κύριος Κιμπαρόπουλος. Από το ΕΛΚ. Έχει τώρα. Έχετε μόνο ένα λεπτό, λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ να είστε ακριβείς με το χρόνο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί Επίτροποι Ντάλι, αγαπητοί συνάδελφοι. Μαχόμαστε όλοι υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων με απειρία ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης τους και είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποιες ε, ψυχικές ή πνευματικές αναπηρίες. Δυστυχώς ο μιλητής είναι ακατάληπτος. Ε, νομίζω ότι τις ε, την κατάσταση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να έχουμε ένα πλήρες πλαίσιο, αλλά μας ανησυχεί το πώς θα συνεχιστεί αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Μπίσοφ, S&D. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητή Κατρίν, ε, αγαπητή Επίτροπε, ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Αναφέρθηκε ήδη αυτό το χάσμα μεταξύ της πραγματικότητας και των υψηλών προσδοκιών μας και επομένως έχω δύο ερωτήσεις. Το, η πρώτη είναι πολύ σημαντική για μένα. Το κεφάλαιο απασχόλησης και ιδιαίτερα των κατώτων μισθών. Η πραγματικότητα παραμένει όπου δεν έχουμε εξασφαλίσει το μισθό, έχουμε τεράστιες εξαιρέσεις στα πλαίσια διαφόρων εργαστηρίων. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουμε, γιατί έχουμε ήδη δει την πρόταση της Επιτροπής για τον τον μισθό και αυτές οι εξαιρέσεις ακόμα εξακολουθούν να υφίστανται. Δεύτερη ερώτηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανείς γιατί έχουμε τόσο πολλά έχουμε τόσο σημαντική πρόοδο παντού, αλλά με την κάρτα αναπηρίας για τους πολίτες ακόμα δεν έχουμε ομοιογενή εφαρμογή. Δεν έχουμε υλοποίηση από τα κράτη-μέλη. Επομένως, κυρία Επιτρόπε, πότε θα έλεγατε ότι πρέπει να έχουμε στα κράτη-μέλη την ίδια κάρτα χωρίς διακρίση σε όλο το έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Την κυρία Μπίσοφ λέει Πρόεδρος. Η κυρία Αλσαλάνη από το Renew, παρακαλώ. Δεν έχουμε σύνδεση, λέει η γραμματεία. Συνεχίζω με το ECR. Ο κύριος Καλησπέρα. Με ακούτε? Πολύ κακά ακούγεται ο κύριος Γκόκκιν. Πάρα πολύ άσχημα. Ακούγομαι. Ναι, σας βλέπουμε, λέει ο συντονιστής. Ναι, με βλέπετε, μ' ακούτε κιόλας όμως. Hello, μ' ακούτε. Ναι, σας ακούμε, λέει ο συντονιστής. Ωραία, ευχαριστώ. Καταρχάς, λοιπόν, ε, να ευχαριστήσω για την ε, έκθεση. Είναι αυτονόητο ότι οι άνθρωποι με αναπηρία ανήκουν ε, στην πολυμορφία και εκφράζουν την πολυμορφία της ε, κοινωνίας. Σίγουρα υπάρχουν ε, κάποια πλαίσια τα οποία πρέπει να ισχύουν για την εκπαίδευση, για την ελευθερία, τη δυνατότητα κινητικότητας, την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία αυτές τις ε, τα συστήματα τα οποία έχουμε για άτομα με αναπηρία, κάποιες ε, κινητές μονάδες ε, για τα άτομα μπορούσε να εφαρμοστεί. Δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά αν θέλουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθήσουμε και αυτές τις... Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τζέμα είναι ο τελευταίος ομιλητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γνωρίζουμε καλά ότι η οδηγία για την ίση μεταχείριση ε, σε θέματα απασχόλησης μόνο μερικώς ευθυγραμμίζεται προς τα Ηνωμένα Έθνη. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι με αναπηρίε εξακολουθούν να υφίστονται περιορισμού των δικαιωμάτων τους, μεταξύ των οποίων την ίση πρόσβαση στην απασχόληση. Επομένως θα πρέπει να ενσωματώσουμε απολύτως τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών στο νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε στα εργασιακά. Επίσης ήθελα να υπογραμμίσω ε, το θέμα των διακρίσεων μεταξύ των φίλων που έχει πολύ ε, ισχυρό αντίκτυπο, μάλιστα πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο, εκθετικό. Κατά των γυναικών που αντιμετωπίζουν αναπηρίες που περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και τα βιολογικά τους δικαιώματα. Ε, πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε τέτοιες ε, ελλείψεις και τέτοια προβλήματα ε, απολύτως επιγόντως. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ντάλη τώρα. Για τις απαντήσεις ελπίζω να είναι ακόμα μαζί μας η Επίτροπος. Έχετε πέντε λεπτά, λέει ο Πρόεδρος, για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε. Λοιπόν, για τους κατώτατους μισθούς. Βεβαίως και αυτό είναι δικαίωμα και θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Θα έλεγα χωρίς καμία εξαίρεση. Βεβαίως και πρέπει να το επιβάλλουμε. Η κάρτα αναπηρίας ε, βλέπουμε απολύτως τις ε, τα ωφέλη της ε, και εξετάζουμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε την εφαρμογή της για την εναρμόνιση και τις ε, ενισχύσεις, τα επιδόματα θα πρέπει να, εδώ να πω ότι πρέπει να σεβαστεί κανείς και το πλαίσιο αρμοδιοτήτων που υπάρχουν. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι απολύτως ε, ενωσιακής αρμοδιότητας. Γνωρίζετε ότι έχω δεσμευτεί να παραδώσουμε μια στρατηγική ώστε τα δικαιώματα που εγγράφονται στις συνθήκες και στη χάρτα να αποτυπώνονται σε υπηρεσίες που θα παρέχονται σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως έχω εξηγήσει τους τελευταίους μήνες, έχουμε πραγματοποιήσει εξαιρετικά εκτεταμένες ε, διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους φορείς και τα κράτη-μέλη και το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο θα συζητηθεί το θέμα των αναπηριών. Η προσωπική μου φιλοδοξία είναι η νέα στρατηγική για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες να έχει αποφασιστικό αντίκτυπο επί της κατάστασης στην απασχόληση και της ευζοίας των ανθρώπων με αναπηρία. Θα πρέπει να αυξήσουμε την συμμετοχή στην αγορά απασχόλησης των ανθρώπων με αναπηρίες, ώστε να κλείσουμε το χάσμα και μεταξύ των φύλων και μεταξύ διαφόρων ευάλωτων ομάδων. Θα πρέπει να μην εκμεταλλεύεται η αγορά το οποιοδήποτε μειονέκτημα που αντιμετωπίζει ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με αναπηρίες, και να τους προστατεύουμε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη μετακίνησή τους και επίσης θα πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους με αναπηρίες από διακρίσεις. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της υιοθέτηση της οριζόντιας οδηγίας κατά διακρίσεων στα πλαίσια της υφιστάμενης οδηγίας κατά διακρίσεων για την προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής ζωής. για διάφορα οριζόντια θέματα για την καλή παρακολούθηση της υλοποίησης της στρατηγικής, για τη συστηματική συλλογή των δεδομένων και ποιοτικών και ποσοτικών. Όλα αυτά είναι κρίσιμη σημασία. Οι ευρωπαϊκοί πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμμορφούμενοι προς το EU CRPD. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση επίσης, που σημαίνει καλύτερη συνεργασία με τους ε, ευρωπαϊκούς, ε, με τους ενωσιακούς θεσμούς, μεταξύ δηλαδή και Συμβουλίου και Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να ηγηθούν ως παραδείγματα στην υλοποίηση EURCPD. Και χρειαζόμαστε ε, συνεχιζόμενη στενή συνεργασία και διάλογο για όλες τις πολιτικές και τα μέτρα που αφορούν στην προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες. Έχω σημειώσει τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις σας και σας βεβαιώ ότι θα διαμορφώσουν, θα αποτυπωθούν στη στρατηγική την, ε, ε, μετά το 2020. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Τώρα για καταλεκτικά σχόλια θα επαστρέψουμε στην κυρία Λάγκεντζη, ε, την εισηγήτρια. Παρακαλώ. Ε, αγαπητή Έλενα, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που ακούσατε τις προτάσεις μας. Ε, χαίρομαι που ακούω ότι η στρατηγική αυτή μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές. Στα πλαίσια της συζήτησης αυτής ήθελα να πω έχοντας υπάρξει νεαρό κορίτσι που, με αναπηρίες, ε, σας βεβαιώνω ότι ε, οι άνθρωποι με αναπηρίες υποφέρουν αλλά δεν υποφέρουν μόνο σωματικά αν θέλετε ή ψυχικά είναι θέμα πλήρους συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθε Πρόκειται για ένα θεμελιώδες και βασικότατο ανθρώπινο δικαίωμα και ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, που μίλησαν, που υπέβαλαν προτάσεις τροπολογιών. Έχουμε προετοιμάσει 35 ε, τροπολογίες ε, συμβαστικές, τις οποίες θα διαβιβάσουμε. Είμαι πολύ θετική για την έκθεση. Προφανώς και εδώ και εκεί ίσως να έχουμε ερωτήσεις, απορίες, προτάσεις βελτίωσης, πράγματα που θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω, αλλά είμαι αισιόδοξη ότι η έκθεση αυτή θα είναι εξαιρετική. Σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά. Για την υποστήριξή σας, αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητή Έλενα, πρόεδρε, ευχαριστώ. Λέει πρόεδρος, ευχαριστώ όλους. Έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή ημερησία διάταξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, γραμματεία, τους τεχνικούς, τους διερμηνείς, όλους αυτούς που συνέβαλαν στο να μπορέσουμε σήμερα να συνεδριάσουμε, να μιλήσουμε. Επόμενη συνεδρίαση 30 Νοεμβρίου στις 4 ε, και 45 εδώ στις Βρυξέλλες το απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.